Well, hello Καλησπέρα. Να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Μερικοί από εσά χάσατε την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους βιώσιμους στόχους ανάπτυξης. Θα μπορούσατε να έχετε μάθει ότι στην ουσία δουλεύουμε στο βρόντο, γιατί η δράση το περιβάλλον είναι κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί. Κρίμα πραγματικά που δεν ήσασταν εδώ για να ενημερωθείτε για το, τα πεπραγμένα μας στην επιτροπή αυτή τα τελευταία πέντε χρόνια. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή τροφή για σκέψη. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία και ας προσπαθήσουμε να εγκρίνουμε την πρόταση για ψήφισμα ε, σε τη φορά την πορτοβουλία για τους επικονιαστές. Ξεκινάμε με την συμβαστική πρόταση 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τροπολογία 50, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49. Τροπολογία ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 64 παρακαλώ, 64, για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 64, αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έχετε δίκιο με μεγάλη πλειοψηφία. Λάθος μου. Να κρίνω μόνο από την δεσκομένα χέρια. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική πρόταση 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100, 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά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 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 109 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά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 τα αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά. Για να ελέγξουμε τη 15 αρχίζει η ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται με δύο ψήφους υπέρ, ε, 16 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται 18 υπέρ κατά Αποχέ αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 19 αρχίζει η ψηφοφορία είναι γλωσσική αυτή η τροπολογία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με μια ψηφοδιαφορά 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 34 υπέρ, κατά αποχές για να ελέγξουμε την 34, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφους. 35 υπέρ κατά, αποχές, μισό λεπτό να το ΕΛΚ, δεν είδα, είστε υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. I want to say hello to Θα καλωσορίσω και μία, και μία ομάδα καλεσμένων ε, και να σας ενημερώσω ότι εγκρίθηκε η πρόταση αυτή. Έχουμε μία ομάδα καλεσμένων από το Χάγκελο των κατοχωρών. Καλώς ήρθατε, ελπίζω να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 την τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος και εγκρίνεται. 27. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ, κατά, αποχές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 κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ένα σχέδιο ψηφίσματος ε, για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία και φροντίδα, στην ενιαία ψηφιακή αγορά, ενισχύοντα τους πολίτες και δημιουργώντας μια γέστερη κοινωνία. Περνάμε στην 32 υπέρ, κατά, αποχές, το ΕΛΚ είναι υπέρ, άρα εγκρίνεται η 32. 33 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά. Αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ, 62 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. And it is closed. And it is adopted. Εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά Tensions. Adopted. Εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ. Καταπίπτει. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 72. You are voting uh, crosswords, so yeah, it's closed. It is adopted. Εγκρίνεται. 74. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά Α, το 94 έχει αποσυρθεί. Μπέλετ, ε, κύριε Μπέλετ, έχω ένα W, άρα έχει αποσυρθεί. 95, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 και 106 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ ή μάλλον καταπίπτει το 10 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά το έλκυνη υπέρ άρα εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 16 άρχεται η ψηφοφορία And is closed. Oh. Τέλος ψηφοφορίας. ισοψηφία. Αυτός που κράτησε απόχη θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται τελικά. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το 23 άρχιτη ψηφοφορία uh, and and it is adopted. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά Το ΕΣΥΑΡΤΗ ψηφίζει και υπέρ και κατά. Α, κατά. Άρα απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. έρχεται η ψηφοφορία. Α. Oh. It is... The vote is closed and it is rejected. Ωραία. Δεν ήταν καν οριακό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Δεν τα είδα καλά. 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά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 Τέλος. Εγκρίνεται τελικά. ολοκληρώσουμε τις ψηφοφορίες. Έχουμε την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση για την εφαρμογή των νομικών διατάξεων Κοινοβουλευτικό ελέγχου σε αποκεντρωμένου οργανισμού και ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι εκπομπέ τη αεροπορία πλην του διοξιδίου του άνθρακα. Και μην ξεχνάτε το ραντεβού μα στι 5 η ώρα που θα έρθει ο Διευθυντή τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, ο Δόκτωρ Γκεμπρεγέσου, που θα μα παρουσιάσει το, παγκο... το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράση για την Υγεία τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Θα ακολουθήσει μνή δεξίωση έξω από την αίθουσα. I insist. Περνάμε στο επόμενο σημείο, που σας είπα. Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινή δήλωση που εξασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, για την οποία η είναι ο κύριος Μπέλετ που έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για τη βραχνάδα στη φωνή, είμαι λίγο κρυωμένος. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων πράγματι εξετάζει την κοινή δήλωση για τις νομικές ε, διατάξεις ε, σχετικά για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, των οργανισμών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας, γιατί είναι αρμόδια για πέντε τέτοιους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Τον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, ΕΚΑ δηλαδή, Περιβαλλοντικό Οργανισμό EEA, Οργανισμό Φαρμάκων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης ε, Ασθενειών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων. Όλοι αυτοί οι πέντε οργανισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των οργανισμών αυτών ε, επίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό να καταρτήσουμε μία γνωμοδότηση και να τη στείλουμε στους συναδελφούς της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων έχουν συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το έλεγχο των αποκεντρωμένων οργανισμών από τι ε, υπόλοιπε ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου. Μπορώ να σας δώσω τις ε, λεπτομέρειες. συζητή είναι ο κύριο Σόπφλιν. Η έκθεση αυτή αναλύει τις εκείνες δηλώσεις από το 2012, δηλαδή έξι χρόνια πριν. Εξετάζει το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί αυτοί και τις συστάσεις για ενδεχόμενη μελλοντική αναθεώρηση της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου των οργανισμών αυτών και ε, της, ε, του συνεχιζόμενου νομοθετικού έργου. Μη, αναφέρομαι στην νομοθεσία για τα τρόφιμα, την έκθεση Ζόμερ δηλαδή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος εστίασα στα θέματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας, αλλά και στις δημοσιονομικές πτυχές, τις οποίες θα επανέλθω συνέχεια κοινοβουλευτικό έλεγχος σημαίνει διακυβέρνηση και διαχείριση του ε, Διοικητικού Συμβουλίου αυτών των οργανισμών. Υπάρχουν εκπρόσωποι από το Κοινοβούλιο, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στα Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και στον έλεγχο των οργανισμών αυτών. Υπάρχουν εκπρόσωποι σε τέσσερις από τους πέντε οργανισμούς, εκτός από τον ΕΦΣΑ, τον ε, Οργανισμό Επιστημιστικής Ασφάλειας, Ασφάλειας των Τροφίμων. Εκεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από την, Επιτροπή, ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως και αυτό βρίσκεται υπό εξέταση στην έκθεση Ζόμερ. Υπάρχει ειδικό σημείο που αναφέρεται ακριβώς στον Οργανισμό Ασφαλής των Τροφίμων. Το σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρομαι στην άποψή μα ότι δηλαδή η κοινή δήλωση του 2012 δεν θα πρέπει να καταδεικνύει πόσα μέλη θα έχει τη δυνατότητα να διορίζει το Κοινοβούλιο στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Αναφέρεται στη γνωμοδότηση ότι χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στην λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και φυσικά ε, πως πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του οργανισμού για τον οποίο είμαστε υπεύθυνοι. Επίσης, στο σχέδιο γνωμοδότησης αναφέρουμε ρητά ότι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ότι δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποδεικνύει στο Κοινοβούλιο πόσους ε, εκπροσώπους θα διορίζει στα Διοικητικά Συμβούλια. Μετά, πρώτο λοιπόν θέμα ήταν η διαχείριση και η διακυβέρνηση και δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η τοποθεσία. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ιδιαίτερα με τον πρώτο. Ε, είχαμε μεγάλα θέματα, διότι φυσικά έπρεπε να μετακομίσει από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ. Ε, γνωρίζετε όλοι τι έγινε, το Κοινοβούλιο δεν ε, συμμετείχε στην διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να καταστήσω σαφές ότι ε, ο τρόπος δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ο συνάδελφος κύριος Λαβία έχει καταρτήσει έκθεση για το θέμα αυτό και εμείς ε, στην ουσία αντιγράψαμε τα όσα αναφέρει στην έκθεσή του και τα χρησιμοποιούμε στην γνωμοδότησή μας. Στην έκθεση Λαβία εκφράζουμε τη λύπη μας ε, για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ε, εκπρόσωποι των πολιτών δηλαδή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτό ψηφίστηκε και στην Ολομέλεια. Επίσης, αναφερόμαστε στη, στο δικαίωμα συμμετοχή στις σημαντικές αποφάσεις, όπως ε, μεταφορά έδραση ή επιλογή έδρας διαφορών αποκεντρωμένων οργανισμών. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στην ε, συνήθη νομοθετική διαδικασία, διότι το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Αναφερόμαστε λοιπόν στην διαδικασία που ακολουθήθηκε έτσι ώστε να επιλεγεί έδρα του, της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και αναφερόμαστε στο ότι στερήθηκε το Κοινοβούλιο των δικαιωμάτων του. Αναφερόμαστε στην έκθεση του 2012, στην κοινή δήλωση. όπου Αναφέρεται σαφώς ότι το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή της έδρας των οργανισμών αυτών. Από την άλλη όμως, η κοινή δήλωση αναφέρει εξίσου σαφώς ότι αυτό δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Επιμένουμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακολουθείτε η διαδικασία για την ε, έδρα των ε, αποκεντρωμένων αυτών οργανισμών. Αναφέρουμε επίσης ότι χρειάζεται αναθεώρηση έτσι ώστε στο μέλλον να μην σημειώνονται τέτοια περιστατικά. Να προσθέσω επίσης ότι ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τονίζουμε αυτό, μέχρι τον Απρίλιο του 2019 να παράσχει μία ενδελεχή ανάλυση της ε, προσέγγισης που ακολουθεί για την επιλογή της έδρας των αποκεντρωμένων οργανισμών, έτσι ώστε να μας οδηγήσει αυτό σε μια νέα συμφωνία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο. Αναφέρουμε επίσης πώς αναμένουμε να γίνονται απόλυτα σεβαστές οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Και όπως αναφέρεται στην έκθεση Λαβία, την οποία υπερψηφίσαμε στην Ολομέλεια πριν από λίγες εβδομάδες, πως είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος των ε, οργανισμών αυτών. Τρίτον, πέρα από την διαχείριση και την ε, έδρα των οργανισμών αυτών, αναφερόμαστε και στη σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό εντάξει είναι λίγο πολύ αυτονόητο. Διότι όταν γίνεται λόγο για τον έλεγχο και το Διοικητικό Συμβούλιο, εξυπακούονται αυτά. Υπάρχει κοινή δήλωση του 2012, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μπούσουλα για να ενισχύσουμε και να ευθυγραμμίσουμε τους ε, μηχανισμούς αντιμετώπισης ε, περιπτώσεων τέτοιων σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν το Κοινοβούλιο εκπροσωπείτε πρέπει να ασχολείται και με τέτοιες περιπτώσεις ε, σύγκρουσης συμφερόντων και να τις αποφεύγει. Η κοινή δήλωση Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθούν και να αυθυγραμμιστούν οι τρόποι πρόληψης τέτοιων περιπτώσεων. Μετά, δεν αναφερόμαστε στους οργανισμούς καθ' αυτούς, χωρίς να μιλήσουμε και για τον προϋπολογισμό. Φυσικά, πάντα στο πλαίσιο του επόμενου πουδουπού, είναι επομένως αναπόφευκτο να αναφερθούμε σε αυτό. Αναφερόμαστε στους δημοσιονομικούς περιορισμούς, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υποκεντρωμένοι οργανισμοί. Αναφερόμαστε επίσης και στις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού και τον μεγάλο όγκο ε, δουλειάς που έχουν να διεκπαιρεώσουν. διότι ο προπολογισμό ε, έχει άμεσες επιπτώσεις ε, στην λειτουργία ενός οργανισμού. Θεωρούμε λοιπόν πως σωστά συμπεριλαμβάνεται και τονίζεται η διάσταση αυτή στην νομοδότηση. Τέλος, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην γνωμοδότηση τονίζουμε την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον, το κλίμα και οι στόχοι μας για το κλίμα στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο Αναφερόμαστε και συγκεκριμένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο οποίος θα αναλάβει πρόσθετες αρμοδιότητες με το νέο πολιτισμο-οικονομικό πλαίσιο. Αναφέρομαστε λοιπόν στον προϋπολογισμό για, όλες τις, για όλους τους πέντε οργανισμούς, ειδικά όμως για τον τελευταίο, τον ε, Οργανισμό Περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν συνοπτικά ήταν τα κύρια στοιχεία της νομοδότησης που θα στείλουμε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Φυσικά είμαι ανοιχτό σε σχόλια και προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Α, να δώσω το λόγο στις, ε, στους σκιώδεις συζητητές. Η κυρία... Η κυρία Μπίλιανα Μπόρζαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Μπέλετ για την πολύ αξιόλογη ε, γνωμοδότησή του. Συμφωνώ και με την προσέγγιση του και με τις απόψεις του. Ε, σε περίπτωση μετεγκατάστασης ε, ε οργανισμών όπως έγινε με τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, ανέκυψαν κάποια προβλήματα που υπάρχουν στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων δύο θεσμικών οργάνων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε και η τελική ε, απόφαση που ουσιαστικά ήταν σαν να ρίχνουμε το κέρμα ε, δεν περιποιεί τιμή στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και μάλιστα μήνες ε, πριν από την ψηφοφορία έγινε γνωστή τελικά ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί. Και μάλιστα τον, τον, τον Ιούνιο ε, ελήφθη η απόφαση και η ψηφοφορία έγινε στα τέλη του, στα τέλη του έτους. Έπρεπε να είχαμε διαμαρτυρηθεί πολύ νωρίτερα. Βέβαια, καλό αργά παρά ποτέ. Έστω και αργά αντιδράσαμε. Και στο τριμερή διάλογο για τη μετεγκατάσταση των δύο οργανισμών, δεχτήκαμε τη διαβεβαίωση ότι στην περίπτωση αυτή είχαμε έκτακτε περιστάσει και στο μέλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί τέτοια διαδικασία όπω αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Στο μέλλον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει από την αρχή τη διαδικασία σε περίπτωση μετεγκατάσταση οργανισμού. Και αν διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα παίρνουν στραβό δρόμο, θα πρέπει αμέσω να αντιδράσουμε. Και η αρχή της γεωγραφικής κατανομής και η με κατάσταση στις νέες χώρες ε, δυστυχώς δεν τηρήθηκαν. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Και η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν αρκετές, αρκετούς οργανισμούς στο έδαφος τους, ενώ πολλές χώρες δεν φιλοξενούν στην επικράτειά τους ούτε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Επίσης, ε, και σε άλλους τομείς θα πρέπει να αναλύσουμε την κοινή δήλωση και το πώς εφαρμόζεται. Και γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω ε, τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τον επόμενο Απρίλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας ε, επισήμανε κάποια θέματα που με βρίσκουν ε, σύμφωνοι. Αναφέρθηκε και επέμεινε στο θέμα ε, της έδρας ε, των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Και αυτό το λέει στο, στα σημεία 2, 3 και 4, στο επίκεντρο δηλαδή της γνωμοδότησης. Και μάλιστα με τις διαπραγματεύσεις του Brexit και με την όλη κατάσταση είδαμε κατάματα την πραγματικότητα και τις φοβερές δυσλειτουργίες που υπάρχουν σε θέματα και οργανισμών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκε πρωτοτελεσμένο γεγονότος και ουσιαστικά έχουμε ένα εξάμεινο που το Συμβούλιο πήρε ομήρους ε, τις, ε, τους οργανισμούς και κυρίως το προσωπικό που βρέθηκε στα διασταυρώμενα πυρά σε αυτή τη διαδικασία. Ε, και έτσι εφαρμόστηκε μια κακή διακασία για τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και αναφέρθηκε ειλικρινή και διαφανή συνεργασία στο κείμενο τη κοινή δήλωση που κανονικά ε, προβλέπεται στην κοινή αυτή δήλωση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Και ουσιαστικά αυτή η κοινή δήλωση έριξε λάδι στη φωτιά, γιατί εμείς ουσιαστικά σκάψαμε το λάκκο μας και για να παραφράσω αυτά που είπε πριν από λίγο η κυρία Μπόρζαν, όλη αυτή η διαδικασία, όλη ε, η ιστορία έγινε για μας ε, το χρονικό ε, μιας προαναγγελθήσης ήτας. Και οι διαπραγματεύσει που, που συνεχίστηκαν στον τριμερή διάλογο οδήγησαν σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τη φορά τη μετακατάσταση των δύο οργανισμών. Και φυσικά τα καταγγέλουμε όλα αυτά και εκφράζουμε τη λύπη μας στη γνωμοδότηση και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ανάλυση αυτού του διοργανικού Μέκου μέχρι τον Απρίλιο, το επόμενο τους, προκειμένου να αναθεωρηθεί. Βέβαια αυτή ήταν μία ε, ελάχιστη ε, λύση που βρήκαμε με το Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική έδρα των οργανισμών και είναι η νιωστή ανάλυση γιατί είχε προβλεφθεί αντίστοιχη ανάλυση και το 2013 και το 2014. Τι θα πούμε και πάλι, τι καινούριο θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη φορά. Ε, γιατί επανειλημμένως ζητήσαμε όχι αναθεώρηση, αλλά πλήρη αναδιατύπωση αυτής της κοινή δήλωσης και να αναγκάσουμε το Συμβούλιο επιτέλους να σεβαστεί τις συνθήκες, γιατί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και δεν θα πρέπει να παραγωνίζεται. Δεν χρειαζόμαστε μία ανάλυση απλώς. Χρειαζόμαστε ρηξικέλευθη αναθεώρηση και το Συμβούλιο θα πρέπει ε, αντί να χρησιμοποιεί το χρόνο και να κολυσιεργεί και να ε, αναβάλει για το μέλλον την ουσιαστική συζήτηση πολλαπλασιάζοντας τα αιτήματα και αναλύσεις δεν μας οδηγεί πουθενά. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί άρδιν αυτή η διαδικασία και από το Συμβούλιο. Έπρεπε να είμαστε πιο αποφασιστική και ελπίζω να μην μείνουν όλα αυτά στο επίπεδο ευσεβών πόθων. Γιατί αν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει να τηρήσει εκείνο τη συνθήκε, θα πρέπει εμεί να το φέρουμε πρώτον ευθυνών. Το ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους ε, Βέλγους συναδέλφους για το δυναμισμό τους. Ευχαριστώ την κυρία για το δυναμισμό της. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς ε, να παραβλέψει. Υπάρχουν άλλα μέλη που θα ήθελαν να πάρουν ε, το λόγο. Η κυρία Γκροστέτ είπε ότι θα ήθελε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς συμφωνώ ε, με τον κύριο Μπελέτση ιδιαίτερα σε ό,τι φορά το θέμα της διακυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση του ΕΟΦ, γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά, είναι αλήθεια ότι αυτή η διαδικασία μας εξέπληξε πραγματικά. Έχουμε την αίσθηση ότι ρυθμίστηκε το θέμα μεταξύ κρατών μελών και ότι το Κοινοβούλιο θα είχε άποψη, αλλά ήταν πάρα πολύ αργά πλέον. Ιδιαίτερα λυπηρό αυτό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για το μέλλον. Τώρα, πιο γενικά, Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και οργάνωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες μετεγκατάστασης των οργανισμών. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που μίλησαν για γεωγραφική κατανομή. Δεν νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Χρειάζονται συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου οργανισμού, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του, ανάλογα με τα ε, συμφέροντά τους. Αυτά δεν αποφασίζονται μέσα από μία ε, ε, αδιαφανή διαπραγμάτευση. Τα κριτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο γεωγραφικός ε, καταμερισμός δεν είναι η καλύτερη λύση. Πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι μία απόφαση που λαμβάνεται προς το κοινωτικό συμφέρον και όχι για το κυβερνητικό συμφέρον. Τώρα, Πέρα από τη μετακατάσταση, ο πολιτικός και δημοκρατικός έλεγχος αυτών των οργανισμών είναι ένα θέμα κομβική σημασία. Αυξήθηκε ο ρυθμός του, αυξήθηκε ε, η ε, ε, συνεργασία του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας και εκεί ακριβώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκήσει την δυνατότητα ελέγχου που έχει οι, μόνο έτσι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να τύχουν της εμπιστοσύνη των συμπολιτών. Γιατί δυστυχώ για ορισμένους, ορισμένες, για ορισμένους οργανισμούς αυτή η ε, εμπιστοσύνη των πολιτών είναι νεκρό γράμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Κάποιος άλλος που θα να πάρει το λόγο για το θέμα. Όχι η Επιτροπή τότε. Κύριε Κλάους, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε μερικά από τα σημεία που έστειξε ο συγητής και άλλα μέρη της Επιτροπής. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Η Επιτροπή, δίχως άλλο, θεωρεί ότι η κοινή προσέγγιση συνεχίζει να παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τους οργανισμούς. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ανάγκη για αναθεώρηση αυτής της κοινή προσέγγισης. Σε ό,τι αφορά το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους διάφορους οργανισμούς και το θέμα του Κοινοβουλίου που εκπροσωπείται συστηματικά στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το Κοινοβούλιο έχει διάφορα μέσα προκειμένου να ασκήσει έναν ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικό έλεγχο, ξεκινώντας με τη διαδικασία του προπολογισμού, αλλά και με τη διαδικασία απαλλαγής και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καλέσει τους διευθυντές ενός οργανισμού σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και να ε, ενημερωθεί για οποιοδήποτε θέμα τον ενδιαφέρει. Η κοινή προσέγγιση που ανέφερα πράγματι προβλέπει ότι το κοινοβούλιο θα μπορούσε να εκπροσωπείται στο δικό συμβούλιο ενό οργανισμού όταν κρίνεται σκόπιμο. Τι σημαίνει αυτό το where appropriate. Αυτό είναι κάτι που μας το δείχνει το ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Πνευματικής ε, Ιδιοκτησίας του Αλικάντε. Ένας οργανισμός που δεν υπόκειται στη διαδικασία απαλλαγή του Κοινοβουλίου και εκεί σαφώς υπάρχει ανάγκη από το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα για να ασκήσει έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάνατε διάφορα σχόλια σχετικά με τη διαδικασία, με την κατάσταση. Καταρχάς, η Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερα που υπάρχει πλήρης νομικής σαφήνεια για την οργανισμό και το προσωπικό. Η Επιτροπή βεβαίως γνωρίζει το την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρξει αυτή η έκθεση για την ε, κοινή προσέγγιση. Η Επιτροπή θα το κάνει αυτό. Μερικοί από εσά ανέφεραν ότι αυτό είναι μια περιγραφή του τι έγινε μέχρι τώρα υπάρχει αυτή η αντίβα, αντίφαση μεταξύ του κοινοβουλίου, του κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Εμείς θεωρούμε, ε, το Φούλε θεωρεί ότι είναι δικής, ε, δικό τους προνόμιο το θέμα ε, αφορά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων πληροφοριακά, δεν να σας πω ότι η Επιτροπή αναθεωρεί τον δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς, η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο είδε τι θα υιοθετήσει ε, θα υιοθετηθεί με τη μορφή κατεξουσιοδότηση πράξης. Το θέμα είναι να ενδυναμώσουμε τους υπάρχοντες μηχανισμούς με κανόνους που επεκτείνονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ακόμα και πιο πέρα. Δηλαδή, όταν πρόκειται για προσωπικό που παρέχει ε, υπηρεσίες σε πελάτες, σε οικονομικούς φορείς. Τέλος, ετέθη το θέμα του προϋπολογισμού και το θέμα των κατάλληλων ε, δημοσιονομικών μέσων ε, χρηματοδότησης. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε στις νέες προτάσεις του δημοσιονομικού πλαισίου, το σημείο εκκένησης ε, για τους διάφορους οργανισμού είναι σταθερότητα και σε ονομαστικούς όρους 20-20. Δηλαδή, σε όλους τους οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη ενδιάζουσες περιστάσεις, νέα καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί, νέα νομοθεσία που τίθεται στην εφαρμογή. Θα υπάρξει λοιπόν μία ε, διαφοροποίηση. Η Επιτροπή Ε, αυτό δεν είναι το θέμα, δεν ε, βρίσκεται στο θεματολόγιο μας και νομίζω ότι ήδη αυτό είναι ένα καλό νέο για την χρηματοδότηση των οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψουμε στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπέλετ, ε, για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι υπάρχει γενική συμφωνία σε ό,τι αφορά τα γενικότερα θέματα η συνάντηση της ΑΦΚΟ συμφώνησαν σε ό,τι αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης όπως ε, ε, το βιώσαμε. Ε, δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνεται τυχαία αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να ορίζονται προκειμένου να αποφευθεί η επιστροφή σε μια τέτοια κατάσταση, λυπηρή κατάσταση, όπου τα πάντα αφήνονται στην τύχη. Η κυρία Ρίσα αναφέρει θέτηκε συγκεκριμένα στις κοινέ δηλώσεις που θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν όχι μια αναθεώρηση αλλά ένα, ε, μια σύνταξη από την αρχή. Ε, είπε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ξεκάθαρη γλώσσα. Η κυρία Μπόσαν ανέφερε σε μια, αναφέρθηκε σε μια εντελεχή ανάλυση που, που θα επιθυμούσαμε η Επιτροπή είναι διάμεση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ε, ε, περιμένουμε να γίνει κάτι μέχρι τον Απρίλιο. Δύσκολο βέβαια το έργο της όπως ε, γνωρίζουμε. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι του, ε, δικό του προνόμιο. Εμείς είμαστε συνομοθέτες βρισκόμαστε ε, μπροστά ε, στο, στο Brexit, αυτή είναι μία πραγματικότητα. Εμείς περιμένουμε ε, να υπάρξουν περισσότερες φιλοδοξίες από πλευρά της Επιτροπής. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Περιμένω προσθήκες Σα όσα ήδη αναφέρθηκαν, πιστεύω ότι είναι προς το δικό μας συμφέρον να υπάρξει μια όσο γίνεται ευρύτερη ε, συμφωνία, έτσι ώστε η θέση μας να γίνει όσο γίνεται πιο δυνατή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνεισφορά σας. 22 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Στις 21-22 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Κατόπιν τίματος των Πρασίνων. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις των αεροπορικών μεταφορών ανεξάρτητα από το διοξίδιο του άνθρακα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι μέχρι τις την 1η Ιανουαρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παρουσιάσει μια έκθεση για τις επιπτώσεις ε, του διεξίου του άνθρακα στην αεροπορία και προτάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις. Ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να Αναθεώρηση Υπάρχει και η έκθεση Girling πάνω στον κανονισμό 2392 του 2017. Έχουμε λοιπόν καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακούσουμε την δική της άποψη και έπειτα τα μέλη της Επιτροπής θα λάβουν το λόγο. Η κυρία Ντίας Πολίτο είναι, θα μιλήσει εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δίνει αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Φλόρες Πολίδο, επικεφαλής έτοιματος ε, αεροπορία στην ε, Γενική Διεύθυνση MOVE. Ανέλαβα τα καθήκοντα σε αυτή τη θέση πριν από λίγους μήνες, γι' αυτό λοιπόν είναι πρώτη φορά που έρχομαι. Και μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω τα, ε, την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να πω ότι θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε στο μέλλον, μια που θα είμαι η αρμόδια για περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα της αερο, των αερομεταφορών. Χθες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Επίτροπό μας ε, στο θέμα του Κορσία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω θυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ε, συμπεριλαμβάνεται και η ε, αεροπλοεία στο πρόγραμμα της Επιτροπής υπάρχει, συμπεριλήφθηκε στο σύστημα πορείας εκπομπών δικαιωμάτων εκπομπών το 2012 και ασκούμε πίεση σε διεθνές επίπεδο για να δημιουργηθούν ε, ισχυροί συμπαγείς κανόνες ε, γι' αυτό. οι εκπομπές ε, της, των αερομεταφορών εκπροσωπούν το 2, ή 3% των συνολικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι όμως οι μόνες εκπομπές που έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή οξυδίων του αζότου ε, είναι, μια από, είναι ένας από αυτούς τους ρήπους, σωματίδια που εκλείονται, ή ε, το διοξίδιο του θείου. Υπάρχουν και άλλες εκπομπές λοιπόν που δεν είναι διοξίδιο του άνθρακα αλλά είναι εξίσου βλαβερές και είναι στο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα, οι εκπομπές αεροπορίας ε, εκπροσωπούν το 2 ή 3%. Να σας υπενθυμίσω μόνο ότι το διοξίδιο του αζότου ε, που εκλείεται από την αεροπορία είναι το 7% των συνολικών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Με, πέρα από το διοξίδιο του άνθρακα και το οξίδιο του αζότου υπάρχουν οι, τα contrails και οι επιπτώσεις τους στο κλίμα. Όμως, ε, αντίθετα με την περίπτωση του διοξιδίου του άνθρακα, τα ίχνη συμπίκνωσης ε, και οι υπόλοιπε εκπομπέ που δεν είναι διοξιδίου του άνθρακα έχουν πτώσει και πρέπει να μειωθούν. Υπάρχει ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα ε, και δεν γνωρίζουμε πολλά. Ε, αβεβαιότητα, τι εννοούμε, τόσο σε κλίμακα, ενώ τον αντίκτυπο, όσο και στο συνολικό πλαίσιο, στις συνολικές εκπομπές. Αυτές οι αβεβαιότητες αυξάνονται ακόμα περισσότερο όταν γίνεται λόγος για τα, τις εκπομπές και τις επιπτώσεις από τα ίχνη συμπίκνωσης. Επιπλέον, δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για την ε, εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Σε ό,τι αφορά το διοξίδιο του αζότου γνωρίζουμε ότι έχει άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ξέρουμε για το διοξίδιο του άνθρακα και το οξίδιο του αζότου ε, πώς μπορούμε να το μειώσουμε. Όμως για τα ίχνη συμπίκνωσης οι γνώσεις μας είναι ελλειπείς. Θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές, αλλά ε, δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα πρέπει να αλλάξει η αεροπορία έτσι ώστε να μειωθούν αυτές οι εκπομπές των ίχνων συμπίκνωσης. Πάνω από 100 χρόνια πετάνε αεροπλάνα, γι' αυτό λοιπόν ε, δεν έχουμε άλλη δικαιολογία και πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές από ίχνη συμπίκνωσης. τα σωματίδια, οξύδια του αζότου, πτυτικές ε, οργανικές ενώσεις είναι, τα είναι σημαντικότερες ενώσεις που εκλείονται από την αεροπορία και δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες ασχολήθηκαν με τον αντίκτυπο των εκπομπών της ε, αεροπλοείας ε, στην... στο περιβάλλον. Επίσης δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες ε, για τις ε, εκπομπές σε μεγάλο υψόμετρο πτήσης. Προσπαθούμε να αναλύσουμε λοιπόν τον συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Πέρυσι ε, στον ΔΟΠΑ εγκρίθηκε μία δέσμη μέτρων, θα τεθεί σε ισχύ το 2020, αναφέρεται στις εκπομπές μη πτυτικών σωματιδίων. Αυτές οι μελέτες έχουν συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία φέτος το Σεπτέμβριο μάλιστα εγκρίθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ. Υπάρχουν πρότυπα τόσο για, τις ε, για τα μη πτυτικά σωματίδια, όσο και για τις εκπομπές που εκλείονται κατά τη ε, διάρκεια της απογειωσής και της προσγείωσης. Αν όλα πάνε καλά, αυτά τα πρότυπα θα εγκριθούν από τον ΔΟΠΑ του χρόνου. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύει εκθέσεις για τις ε, εκπομπές ουσιών εκτός από το διοξίδιο του άνθρακα μέχρι το 2020. Και σας ε, βεβαιώνω ότι κάνουμε ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να τηρήσουμε την υποχρέωσή μας αυτή εγκαίρως. Την έκθεση αυτή, όπως είπα, θα πρέπει να συνοδεύει και μια πρόταση, εφόσον αυτό κριθεί κατάλληλο, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την οδηγία. Ε, και από μένα αυτά προς το παρόν. Περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας και θα σας απαντήσω με μεγάλη μου χαρά πρωτού συνεχίσω. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ποιο ε, ποιος θέλει το λόγο. Έχουμε ήδη δύο μιλητές στο κατάλογο. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι λίγο μπερδεμένο για το ότι έρχεται κάποιο από το Γενική Διεύθυνση MOVE, διότι σύμφωνα με αυτά που ξέρω, η Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο θα έπρεπε να είναι η αρμόδια. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν, ποιο καταρτίζει την έκθεση. Δεν θα έπρεπε να είναι η Γενική Διεύθυνση η οποία ήταν αρμόδια και για τη σχετική νομοθεσία. Ήδη το 2008, όταν είχε ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο αυτό, και το λέω αυτό γιατί ήμουν συγητής της έκθεσης αυτής, γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοιχεία. Ήδη από τότε το ξέραμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν από το 2008 μέχρι σήμερα, αυτά τα 10 χρόνια έχει κάνει κάτι για να αλλάξει ε, αυτό, γιατί διαφορετικά θα πληγεί η αξιοπιστία της. Δεν είναι δυνατόν εδώ και δέκα χρόνια να μας λέτε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Καθυστερούμε, κολλησιεργούμε σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Δεν γίνεται λοιπόν να συνεχίσει αυτό. Ιδιαίτερα στο θέμα της εμπορίας ε, δικαιωμάτων εκπομπών έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Και είδαμε ότι η συμπρόοδο που έχει σημειωθεί δεν είναι επαρκή. Τώρα βλέπω να επαναλαμβάνεται το ίδιο. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να προχωρήσουμε ακόμα και όταν η βάση δεδομένων μας είναι ελλειπής. Δεν νομίζω ότι αυτό το αμφισβητεί κανείς. Μπορούμε να οτικοποιήσουμε κάποια δεδομένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες μελέτες για να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Νομίζω πως ε, εδώ ε, πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Σας ευχαριστώ κύριε Σεκχάουτ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Τουλάχιστον α, σημείωσα ότι πριν την πρώτη η Πρώτου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει την έκθεσή της. Τι έγινε όμως με αυτά που προτείναμε εμείς και τι δράσεις ε, μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκεί ο χρόνος πιέζει και έχω την αίσθηση ότι αυταλαντεύεται κάπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθυστερεί και δεν ξέρω γιατί. Ξέρουμε που έχει φτάσει η επιστήμη και γνωρίζουμε ότι κάποιες τέτοιες ουσίες ε, και σωματίδια επηρεάζουν το κλίμα πολύ περισσότερο από ένα μόριο διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σαφέ ότι επηρεάζουν το κλίμα, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώ, αλλά είναι σαφέ ότι η αεροπορία συνεισφέρει σε αυτόν τον επηρεασμό του κλίματο. Και είναι αδιαφυσβήτητα αυτά τα επιστημονικά πορίσματα και οι συνέπειε αεροπορία στο κλίμα. Τώρα, αν υπενεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρώτα θα πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι για, τις, ε, για το πώ επηρεάζονται τα σύννεφα ε, και ε, ότι τα οξύδια του βρίσκονται μόνο σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ε, ναι, σίγουρα υπάρχει συγκέντρωση οξυδίων του αζότου στις ψηλά, στα υψηλά επίπεδα και σίγουρα επηρεάζεται το κλίμα. Και κοιτάξτε την έκθεση του IPCC για το, την αύξηση του πολύ 1,5 βαθμού. Το IPCC είναι το αρμόδιο και αρμόδιο φορέας του ΟΗΕ για το κλίμα και εκεί αναφέρονται οι ουσίες αυτές που έχουν βραχία ζωή και αν δεν αντιμετωπίσουμε τις ουσίες αυτές, τις βραχύβιες αυτές ε, ουσίες, δεν πρόκειται να τηρήσουμε το στόχο της, μία της πέραν του 1,5 βαθμού Κελσίου. Ε, και μάλιστα δεν μπορούμε να έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα που μιλάει για 1,5 βαθμό και απ' την άλλη να ε, διστάζουμε ε, και να καθυστερούμε για το θέμα αυτών των μη πτυτικών νεωρούμενων σωματιδίων. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των βραχίβιων αυτών ουσιών, αποκλείεται να υλοποιήσουμε το στόχο τη μη αύξηση πέραν του 1,5 βαθμού. Τώρα, ε, στο, ίδιο, στο ίδιο καλάθι ε, διαφορετικά θέματα. Για τα οξύδια του έχουμε ήδη από το, από το 2008 ε, μελέτη που θα πρέπει που λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο παράγων απόσταση για το οξύδιο του αζώτου. Ήδη από το 2008 έχουμε μελέτη και από τότε είχαμε ζητήσει δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα τις περιμένουμε. Δεν διαβάσετε την έκθεση του 2008. Και τι πρόκειται να κάνετε με τις συστάσεις της έκθεσης, γιατί ε, η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική σήμερα και το ζήτημα ακόμη πιο κατεπήγον. Σε ό,τι αφορά τα, τις ουρές συμπυκνώσεις και τα ε, ε, την ε, δημιουργία νεφών, το θέμα είναι τι μέτρα θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτό το γνωρίζουμε και για τα αιρούμενα σωματίδια. Εκεί γνωρίζουμε ότι η αποθειοποίηση της κυροζήνης ε, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Και θέλω συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις επιμέρους ουσίες που γνωρίζουμε ότι θα έχουν συνέπειες. Δεν πρέπει να περιμένουμε τις επιστημονικές μελέτες για τον ακριβή αντίκτυπο, γιατί έτσι θα καθυστερήσουμε πολύ και ξεχάστε τον 1,5 βαθμό Κελσίου που ζητά το IPCC, ο αρμόδιος φορέας του ΙΕ για το κλίμα. Και έχουν περάσει 10 χρόνια από το 2008 που είχαμε την πρώτη μελέτη για το οξύδια του αζότου και τίποτα δεν έγινε στο μεταξύ. Ευχαριστώ κυρία Εκχώτη, κυρία Κούτελαντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και μας παρουσίασε τις απόψεις της και χαίρομαι που υποσχεθήκατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να εκπονήσετε τη μελέτη για τις συνέπειες της αεροπορίας ε, πέραν των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ελπίζω να το κάνετε, ε, γιατί περιμένουμε την έκθεση που την αναγγείλατε για τις αρχές του 2020. Πάντως θα σας πω και εγώ από την ομάδα με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντε, ότι είναι πολύ ανησυχητικό που δεν ακούσαμε περισσότερα για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί έχει περάσει μία δεκαετία. Και ήδη το 2008 είχαμε την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, που αναφερόταν ότι όλες οι συνέπειες της αεροπορίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Και το είδαμε αυτό με την πρόσφατη προειδοποίηση του IPCC. Έκρουσε τον κόδωρο του κινδύνου η ΕΕ και είπε ότι είναι κρίσιμο να λάβουμε υπόψη αυτέ τι ουσίε για να τηρήσουμε τις ε, υποσχέσεις που δώσαμε στο Παρίσι και σίγουρα όλες οι εκπομπές συμβάλλουν στην θέρμανση του πλανήτη. Και δεδομένων των συνεπειών που έχουν ε, εκπομπές αεροπορίας και πέρα του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε κάποια μέτρα και γιατί δεν είχαμε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, με πανεπιστήμια, πανεπιστημιακούς επιστήμονες, με σφαιροντούχους, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία ε, και δεν είναι σοβαρός τρόπος αυτός να καθυστερούμε τόσο πολύ. Επίση, ποια είναι η Γενική Διεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φέρει την ευθύνη για όλα αυτά, γιατί και εδώ υπάρχει ασάφεια. Και συμφωνώ με του συναδέλφου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο ότι δεν είναι σοβαρή αυτή η συμπεριφορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμέναμε πολύ περισσότερα και θα πρέπει τέλο να περάσουμε στα έργα. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι τώρα στην Επιτροπή, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ που μας ξαναδίνετε το λόγο. Θα ήθελα να διαβεβαίωσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή μιλάει με μία και μοναδική φωνή. Ε, Βεβαίω εγώ βρίσκομαι εδώ, δίπλα μου είναι η συνάδελφοί μου τη Γενική Διεύθυνση για το κλίμα. Συνεργαζόμαστε στενά για το σύστημα Κορσία και αυτή η συνεργασία βελτιώνεται κάθε μέρα. Μη φοβάστε το γεγονός ότι ηγείται η DG Lead, δεν σημαίνει ότι δεν εμπλέκεται και η DG Κλίμα και ότι θα αποκλειστεί από τις εργασίες μας. Το αντίθετο. Δεύτερον, Καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το θέμα της αξιοπιστίας, ότι από το 2008 δεν έχει αναφερθεί η Επιτροπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή ε, υπήρξε αδρανής. Καταρχάς έχουμε τις περιβαλλοντικές εκθέσεις που εκδίδονται μαζί με το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο. Η τελευταία εκδόθηκε το 2016, μια άλλη θα εκδοθεί στις αρχές του χρόνου και υπάρχουν βεβαίως εκθέσεις για συγκεκριμένα με, ε, θέματα, το διοξίδιο του θείου και θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον. Δεύτερον, Εκτός από τις εκθέσεις έχουμε το θέμα των αποστολών, συνεργαζόμαστε με την ΔΟΠΑ, με την ΕΑΣΑ προκειμένου να υπάρξουν τα αναγκαία πρότυπα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Ξέρετε ότι καταβάλουμε προτάσεις για περισσότερο βιώσιμα καύσιμα που θα μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρατος. Ξέρετε ότι ότι εργαζόμαστε και με τους ενιαίους ουρανούς για να μπορούν οι πτήσεις να είναι περισσότερο απολετικές. Ξέρουμε ότι έχουν αυξηθεί οι εκπομπές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν κατέβαλε προσπάθεια τομέα των ενέργειων μεταφορών. Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη της αεροπορίας είναι πολύ πιο γρήγορη από την παράλληλα προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές. Εγώ δεν λέω ότι τα θέματα του κλίματος δεν είναι ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή. Λέω ότι μερικές φορές θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα ακόμα και αν προχωράει η τεχνολογία μπορεί αυτό να μην είναι επαρκές. Τώρα για να φερθώ και σε άλλες πρωτοβουλίες. Ξέρετε ότι έχουμε την πρωτοβουλία καθαρή ουρανή για να έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλες οι έρευνες ε, που για την βελτίωση των λειτουργιών και της τεχνολογίας θα φτιάσει μέχρι την αγορά. Η Επιτροπή, η DG Κλίμα, η DG ε, Περιβάλλον έχει αναλάβει δέσμευση έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε θέματα που αφορούν το κλίμα. Καταλαβαίνω βεβαίω ότι θα πρέπει να υποβληθεί η έκθεση σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνω ότι μερικοί από εσά θα ήθελαν να έχουν απαντήσεις σήμερα. Δυστυχώς δεν μπορεί να κάνω κάτι περισσότερο. Εγώ θα πρέπει να πάρω όλη τη βιβλιογραφία. Έγιναν έρευνε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για ε, ορίζοντα 2020 έρευνα, ναι, έγιναν έρευνε παγκοσμίω και εμεί θα πρέπει τι έρευνε αυτέ να τι ε, συγκεντρώσουμε και μόνο μετά από ένα χρόνο θα ξέρουμε πώ ακριβώ έχουν τα πράγματα και πόσο φιλόδοξοι μπορούμε ε, να είμαστε. Αυτό δεν είναι για σήμερα. Θα υπάρξει και μία άλλη ανταλλαγή απόψεων. Εμείς θα επανέλθουμε εδώ για την υποβολή της έκθεσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι είναι πρόωρο το να σκεφτείτε ε, το τι θα κάνει η Επιτροπή με αυτή την ε, πρόταση. Είμαστε το 2018, μιλάμε για ένα ε, νέο κολέγιο επιτρόπων, για ένα νέο κοινοβούλιο. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι πράγματι καταλαβαίνουμε ότι το κοινοβούλιο το 2008 ήθελε τα μέτρα που ετέθησαν επιτάπητος η πλειοψηφία ε, είχαν, έκαναν μία αναφορά στα πρότυπα. Σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, ε, έχουμε κάνει κάτι. Το θέμα των τελών είναι θέμα ε, που ξεφεύγει από τα όρια της Ευρώπης. Θα πρέπει να, έχουμε, να μην έχουμε μια ουτοπική συμπεριφορά σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Εμείς τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη. Σε αυτή όμως τη φάση δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό και μας μένουν δύο λεπτά μέχρι να φτάσει ο κύριος Τάντρος, διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σας παροτρύνω λοιπόν να παραμείνετε στην αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Δ. Τέντρος, ο οποίος εξελέγει Γενικός Διευθυντής για πέντε χρόνια από τα κράτη-μέλη, το Μάιο του 2017. Πριν από την εκλογή του, ο Δ. Τέντρος ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Αιθιοπίας και με την ιδιότητα αυτή ηγήθηκε των προσπαθειών ε, για τη δρομολόγηση του θεματολογίου της Αντίσα Μπέμπα σε 193 χώρες, οι οποίες δεσμεύτηκαν να ε, χορηγήσουν την ε, κατάλληλη χρηματοδότηση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Υπηρέτησε επίσης ως Υπουργό Υγείας της Αιθιοπίας και ήταν επικεφαλής μιας ε, βαθιάς μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας της χώρας. Από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιούλιο του 2017, ο Δόκτωρ Τέντρος υπογράμμισε πέντε μεγάλες προτεραιότητες. Καθολική κάλυψη υγείας, ε, ε, περιπτώσεις έκτακτες ανάγκης στην υγεία, παιδική και εφηβική υγεία, υγεία και περιβαλλοντική αλλαγή και η μεταρρύθμιση του ΠΟΗ. Όπως γνωρίζετε, φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ε, Οικουμενική Διακήρυξη των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ένα έγγραφο ορόσημο το οποίο ενέπνευσε ένα μεγάλο σώμα νομικά δεσμευτικών συνθήκων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε την εξουσία του για να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης και για να ανανεώσουμε την δέσμευσή μας, καθώς επίσης και για να γιορτάσουμε την 70η επέτειο του ΠΟΗ, Δημιουργήσαμε την Εβδομάδα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο τη ε, θα διεξαχθεί σήμερα η σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τον Δόκτωρα Τέντρος. Θα γιορτάσουμε μαζί τα 70 χρόνια πόη. Νωρίτερα σήμερα συζητήσαμε την έκθεση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. και την έκθεση παρακολούθησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018. Είδαμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ο Δ. Τέντρος ε, μου είπε δημερός ότι θέλει να σταθεί σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο θα σας παρουσιάσει στη συνέχεια. Θα περιοριστώ μόνο στο να πω ότι η ανταλλαγή απόψεων θα αποτελέσει ευκαιρία και για εμάς να αφήσουμε ένα κληροδότημα στο επόμενο κοινοβούλιο, να δημιουργήσουμε μία ομάδα σύνδεσης, μία ομάδα φιλίας ανάμεσα στην Επιτροπή μας και ε, στον ΠΟΗ. Με τη βοήθεια του Γενικού του Διευθυντή ελπίζουμε στην επόμενη θητεία να επισημοποιηθεί αυτή η προσπάθεια και να πάρει τη μορφή μιας ε, κανονικής ομάδας. Στο πλαίσιο της ε, συζήτησης θα εξετάσουμε τις λεπτομέρειες αυτής της ε, επιθυμίας μας για στενή συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΠΟΗ και μαζί με τον ε, Δ. Τάντρο θα δημοσιεύσουμε μια κοινή δήλωση η οποία θα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την ε, δημιουργία μιας πραγματική εταιρική σχέσης με στόχο το μέλλον. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστέρηση, δίνω το λόγο στον Δ. Τάντρο. Είναι τιμή μα που σας έχουμε εδώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Βαλεάν, εξοχότητες κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ομίγυρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ, έχω ξανάρθει. Κάτι που δείχνει την ισχυρή εταιρική σχέση και συνεργασία που έχουμε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τελευταίο διήμερο ήταν πολύ καρποφόρο, πολύ επικοδηματικό για την εμβάθυνση των σχέσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα είχαμε σημαντική αύξηση στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ΠΟΕ, ειδικά φέτος, και συμφωνήσαμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας ακόμη περισσότερο. Χθες μίλησα στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και στην ετήσια συνάντησή μας για την έκκλησή μας για να αντιμετωπίσουμε τα έκτακτα περιστατικά, τις έκτακτες ανάγκες. Και μάλιστα συζήτησα αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο Γιούγκερ τον, ε, και τους επιτρόπους ε, Ανδριουκάητης, Μίμητσα, Βέλα και το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Στυλενίδη για την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία για μα. Και όπω ξέρετε, το 2018 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, γιατί εορτάζουμε τα 70 μα γενέθλια. Ταυτόχρονα είναι η 70η επέτειο ε, τη Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και η ίδρυση τη ΠΟΗ και η Οικουμενική Διακήρυξη επιβεβαιώνουν ε, το γεγονός ότι η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι ένα προνόμιο μόνο όσο έχουν τους σπόρους να την αγοράσουν. Και μάλιστα με τον καιρό το δικαίωμα αυτό βρήκε το δρόμο του και μέσω του εθνικού και του διεθνούς δικαίου. Και πολλές χώρες σήμερα έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα στην υγεία στους καταστατικούς τους νόμους, στα συντάγματά τους. Και έχουμε και τρεις διεθνείς ε, συνθήκες για την υγεία. Ε, ε, το σχέδιο σύμβασης για τον έλεγχο ε, του καπνού και την προσπάθεια να απαλληθεί το λαθρομπόριο καπνού και επίσης ε, έχουμε νομικά δεσμευτικές συνθήκες ε, για την υγεία. Είμαστε μάλιστα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ισχυρό υπέρμαχο αυτών των πολυμερών συνδικών και σα ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σα. Βέβαια, το δικαίωμα στην υγεία δεν είναι απλώ μια ευγενή ιδέα ή ένα έγγραφο. Τα τελευταία 70 χρόνια ήταν το εφαλτήριο για σημαντικέ βελτιώσει στην παγκόσμια υγεία. Και από το 1948 το προσδόκιμο ζωή έχει αυξηθεί κατά 25 χρόνια κατά μέσο όρο παγκοσμίω. Η θνησιμότητα των μητέρων και των παιδιών μειώθηκε κατακόρυφα. Η ευλογία έχει εξελιχθεί και η πολιομελίτιδα έχει σχεδόν εξελιχθεί. Και μάλιστα αντιστρέψαμε την αρνητική τάση της επιδημίας του AIDS. Οι θάνατοι από ελονοσία έχουν μειωθεί αισθητά. Τα νέα εμβόλια έχουν κάνει προηγουμένω τρομακτικές ασθένειες αποτρέψιμες πια και υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για να το γιορτάσουμε. Βέβαια, παρόλο που συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τις παλιές απειλές, έχουν ε, αναδειχθεί καινούργιες απειλές. Οι κλιματικές αλλαγές που θα έχει σημαντικές συνέπειες στην υγεία, επίσης η μικροβιακή αντοχή έχει τον, ε, τον κίνδυνο να ακυρώσει τα ωφέλη της σύγχρονης ιατρικής και η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών νέων και μη μεταδοτικέ ασθένειε όπω καρδιακέ παθήσει, κεφαλικά καρκίνο, διαβήτη, υπέρταση, πνευμονοπάθειε και ψυχικά νοσήματα έχουν γίνει βασικοί δολοφόνοι των σύγχρονων καιρών. Και φυσικά συνεχίζουμε να αντιμετωπίσουμε την πανταχού παρουσία των επιδημιών και άλλων έκτακτων περιστατικών. Το Τελευταίου 12 μήνε η ΠΟΗ έχει ανταποκριθεί σε 47 έκτακτε ανάγκε σε 50 χώρε. Και όπω ξέρετε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να περιορίσουμε την επιδημία του έμπολα στην Δημοκρατία του Κονγκό, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουγγάντα. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 366 κρούσματα και 214 θάνατοι από την ε, αρχή της επιδημίας τον Αύγουστο. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να αποτρέψουμε την ε, διασυνοριακή εξάμπλωση του έμπολα, γιατί έχουμε καλύτερα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε το έμπολα, καλύτερα από ποτέ. Και πάνω από 32.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την εξάπλωση της επιδημίας και να κρατήσουμε χαμηλό τον αριθμό των κρουσμάτων Επίσης, έχουμε και ερευνητικέ θεραπευτικές αγωγές ε, για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα κρούσματα. Μέχρι στιγμής 145 άνθρωποι έχουν ε, λάβει θεραπευτική αγωγή με ένα από τα τέσσερα φάρμακα. 14 εκατομμύρια ε, ταξιδιώτες έχουν ελεγχθεί και πάνω από ε, 490 ε, ασφαλείς και αξιοπρεπείς αταφές είχαμε. προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια επαγρύπνηση. Πήγαμε σε 4.000 νοικοκυριά και έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 500 ε, αρχηγούς ε, κοινοτήτων και μάλιστα έχουμε ε, πολύ στενή εταιρική σχέση και πρωτοστατούμε στην ενημέρωση των εταίρων στα θέματα αυτά. Βέβαια, είναι δύσκολο να ελέγξουμε την επιδημία λόγω τη κατάσταση ασφάλεια στο Κονγκό. Ένοπλε δυνάμει που δραστηριοποιούνται στην περιοχή πραγματοποιούν τακτικέ επιθέσει στην πόλη Μπένι, που είναι το επίκεντρο τη επιδημία. Και κάθε φορά που έχουμε μία επίθεση, εποφελείται ο ιός και παρεμποδίζονται τα, ε, οι εμβολιασμοί. Πριν από δύο εβδομάδες πήγα στην Μπένι με τον Ζαν Πιέρ Λακρουά, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατήρηση Ειρήνης και πραγματικά ε, εμψυχώθηκα από τον τρόπο που δουλεύουν τα μέλη του, της οικογένειας του ΟΕΑ. Και μάλιστα την Παρασκευή είχαμε μια επίθεση στο ξενοδοχείο που έμενε το προσωπικό μας και την ώρα που γινόταν η επίθεση ένας υπάλληλό μας που τηλεφώνησε. άκουκα από μακριά τους ε, πυροβολισμούς από το τηλέφωνο, κάτι που σημαίνει ότι ήταν πολύ κοντά στην επίθεση και αργότερα είχα μια κλίση με βίντεο, είδα το φόβο αυτό των ανθρώπων και τους ρώτησα τι θέλετε να κάνετε. Μου είπαν όμως ότι δεν θέλουν να φύγουν, ήθελαν απλώς περισσότερη προστασία για να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να θέσουν ένα τέρμα στην επιδημία του έμπολα. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η διαπίστωση για μένα και καθημερινά νιώθω μεγάλη ταπεινοφροσύνη και ταυτόχρονα μεγάλη έμπνευση από το προσωπικό του ΟΗΕ που θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο για να προστατεύσει το δικαίωμα στην υγεία, για να σώσει ζωές, για να προστατεύσει τους συνανθρώπους μας. Και αυτό μου δίνει εμπιστοσύνη ότι με την υποστήριξη όλων των εταίρων μας θα μπορέσουμε και θα τα καταφέρουμε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την επιδημία. Αλλά όπως έχω πει και επανειλημμένος και θα συνεχίσω να το διατρανώνω, ε, η ασφάλεια της υγείας και τα στήματα υγείας είναι η διόψη του ίδιου νομίσματος. Ε, οι καλύτερες ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πρόθεση και προστασία του δικαιώματος της υγείας είναι η επένδυση σε ισχυρότερα συστήματα υγείας. Η διακήρυξη του Άλμα Άτα πριν από 40 χρόνια εντόπισαν τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας ως το θεμέλιο για την υλοποίηση του δικαιώματος υγείας για όλους. Και μάλιστα είδαμε πως η πολιτική και η οικονομική πραγματικότητα άφησε ανεκπλήρωτο το όραμα του Αλμάτα. Και έτσι στην Αστάνα στο Καζακστάν το περασμένο μήνα συναντηθήκαμε και πάλι για να επιβεβαιώσουμε το όραμα της διακήρυξης ε, του Αλμάτα. Γιατί μόνο με την ε, πρωτοβάθμια παροχή υγείας θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το οικουμενικό δικαίωμα τη υγείας, την καθολική κάλυψη και του ε, στόχου βιώσιμη ανάπτυξη για την υγεία. Και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε αμύωτε τι προσπάθειε μα ε, για την πολιτική δέσμευση. Και επίση ε, ζητούμε από την παγκόσμια κοινότητα να συνεργαστεί με την ΠΟΕ με πιο συνεπή και ολοκληρωμένο τρόπο. Και γι' αυτό η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία και άλλε δέκα διεθνεί υπηρεσίε και οργανισμοί συμφώνησαν να συνεργαστούν σε ένα παγκόσμιο σχέδιο δράση για την υγεία και την ευημερία εγκαινιάσαμε την πρώτη φάση του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης. Σας το έχω φέρει και εδώ, μπορείτε να το κοιτάξετε. Εγκαινιάσαμε λοιπόν αυτή την πρώτη φάση στο Βερολίνο τον περασμένο μήνα και θα παρουσιάσουμε το οριστικό σχέδιο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο του χρόνου κατά την συζήτηση, συνεδρίαση υψηλού επίπεδου για την καθολική κάλυψη υγείας. Και μάλιστα θα ήθελα να ευχαριστήσω την καγκελάριο Μέρκελ που πρωτοστάτησε ε, στις προτάσεις για το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης μαζί με τον Πρωθυπουργό Ζέλμπερ από την Ορβηγία και τον Πρόεδρο της Γκάνα, τον κύριο Άρντο. Το σχέδιο έχει τρεις στρατηγικές προσεγγίσεις. Την ευθυγράμμιση, την επιτάχυνση και τη λογοδοσία. Πρώτον, θα πρέπει να δεσμευτούμε να ευθυγραμμίσουμε πολλέ διαδικασίε μα προκειμένου να αυξήσουμε τη συλλογική μα αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, δεσμευθήκαμε να επιταχύνουμε την πρόοδο εντοπίζοντα ε, τους ε, τομείς ε, εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την καμπή και να κάνουμε πιο ταχεία πρόοδο για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να αφήσουμε την υγεία, όπως ε, έρευνα και ανάπτυξη, δεδομένα και ε, βιώσιμη χρηματοδότηση. Και επίσης θέλουμε να είμαστε υπόλογοι και σε αυτούς που υπηρετούμε και στους ε, εταίρους και δωρητές μας, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, που περιμένουν αποτελέσματα από τους πόρους που μας εμπιστεύονται και που θέλουν να πιάνουν τόπο. Γι' αυτό είπαμε ευθυγράμμιση, επιτάχυνση και λογοδοσία, που είναι τα θεμέλια της νέας, του νέου σχεδίου δράσης. Στα τελική ανάλυση, το μέτρο της επιτυχίας μας δεν είναι ο αριθμός των εκθέσεων που συντάσσουμε, των συνεδριάσεων που οργανώνουμε ή το ποσό που επενδύουμε. Σε τελική ανάλυση, το μέτρο τη επιτυχία μα είναι οι ζωέ που αλλάζουμε. Είναι τα παιδιά που επιβιώνουν και μετά τα πέμπτα του γενέθλια. Είναι οι γυναίκε που θα μπορούν να επιλέγουν κατά πόσο, πότε και με ποιον θα μείνουν έγκυε. Είναι οι άντρε που δεν θα πεθαίνουν πρόωρα από μη μεταδοτικέ ασθένειε. Θα είναι οι οικογένειε, οι κοινότητε και τα έθνη που θα ευδοκιμούν με υγιείς και παραγωγικούς πληθυσμούς. Και όλα αυτά ξεκινάνε με την πεποίθηση ότι η υγεία δεν είναι προνόμιο των ευπόρων, αλλά δικαίωμα όλων. Τα τελευταία όμως 70 χρόνια κατέδειξαν ότι η υγεία για όλους δεν είναι μόνο ένα ευγενές σύνθημα, είναι κάτι το εφικτό. Και αυτό φαίνεται περισσότερο στην Ευρώπη, πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι οι σημεοφόροι του δικαιώματος στην υγεία. Η Ήπειρος αυτή είναι το λίκνο της καθολικής κάλυψης υγείας. Και σκέφτομαι ιδιαίτερο στην Δανία, τη χώρα στην οποία έλαβα την πρώτη ασφάλεια υγείας ως φοιτητή στη δεκαετία του 80. Και μάλιστα αυτή η εμπειρία που είχα τότε άφησε μια ανεξίτηλη μνήμη πάνω μου. Έχουμε πολλά ε, συστήματα υγείας ε, στην Ευρώπη και παροχή οικονομικής προστασίας. Όλα όμως στηρίζονται στο δικαίωμα της υγείας. Πολλές χώρες Ευρώπης ε, δεν δημιούργησαν τα συστήματα υγείας τους όταν ήταν εύπορες. Πολλές ε, τα δημιούργησαν την επαύρη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που οικονομικά ήταν γονατισμένες αυτές οι χώρες. Και μάλιστα αυτό που ισχύει είναι το αντίθετο, ότι οι χώρες αυτές έγιναν ε, σταθερές και ευημέριζαν εν μέρη τουλάχιστον επειδή επένδυσαν στο δικαίωμα στην υγεία. Έκαναν μια πολιτική δέσμευση. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Πολλές άλλες χώρες στον κόσμο, από τη Ρουάντα μέχρι την Ταϊλάνδη και το Περού, που πρόσφατα έκαναν την πολιτική επιλογή να επενδύσουν στο δικαίωμα στην υγεία και να πραγματοποιήσουν πρόοδο. Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας υποβάλω τρία αιτήματα, τρεις εκκλήσεις. Πρώτον, συμφωνούμε ότι η υγεία είναι ένα δικαίωμα σας. Θερμοπαρακαλώ λοιπόν να συνεχίσετε να είστε υπέρμαχοι αυτού του δικαιώματος και οι υπερασπιστέ του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από τα πιο προηγμένα συστήματα υγεία στον κόσμο, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα ισότητα σε κάποιε χώρε. Και φυσικά θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα για να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, κανένα συνανθρωπών μα. Και το συζήτησα με την Πρόεδρο. Το θέμα τη ισότητα, τη ίση πρόσβαση στην υγεία είναι ένα ζήτημα που και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να σημειώσει πρόοδο και συμφωνούμε ως προς την εκτίμηση και την αξιολόγηση. Επίσης, θα ήθελα να σας παροτρύνω να είστε συνήγοροι του δικαιώματος της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό χρειαζόμαστε την πρωτοκαθεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της ηγεσία αλλά και την οικονομική της εμπλοκή. Γιατί χάρη σε παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σώζουμε και παρατείνουμε ζωές. Αλλά προσφέρουμε και πολύ περισσότερα. Βγάζουμε κόσμο από τη φτώχεια, βάζουμε τα θεμέλια της βιώσιμης ανάπτυξης και διαμορφώνουμε την υγιέστερη, ασφαλέστε, τον υγιέστερο, ασφαλέστερο και δικαιότερο κόσμο που όλοι λαχταρούμε. Και τρίτον, σας παροτρύνω να στηρίξετε το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την ε, υγεία και την ευημερία, το έγγραφο που σας παρουσίασα προηγουμένως. Και μάλιστα μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία διαβούλευσης και περιμένουμε τα σχόλιά σας για το πώς μπορούμε όλοι στην παγκόσμια κοινότητα με πιο έξυπνο τρόπο να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και τις επαναλήψεις, να αναβαθμίσουμε την καινοτομία, να την διευρύνουμε. Χρειαζόμαστε νέες ιδέες για κάτι τέτοιο και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω εδώ σήμερα και για τη δέσμευσή σας υπέρ της προστασίας και της προώθησης του δικαιώματος στην υγεία. Ακόμη και σήμερα που εορτάζουμε την 70η επέτειο και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Οικουμενικής Διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το δικαίωμα στην υγεία δεν είναι δεδομένο, δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται πολιτική, ανανεωμένη πολιτική δέσμευση και η ηγεσία σε κάθε γενιά και στη δική μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Καταρχάς, κύριε Γενικέδη Διευθυντή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, προκειμένου να μεταφέρετε ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα γιατί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επικέντρωσε τις προσπάθειές τους θεωρώντας δικαίωμα την πρόσβαση σε υπηρεκίες υγείας. Η κατάσταση βέβαια παραμένει πολύ ανησυχητική και το δικαίωμα στην υγεία πολύ απέχει από το να είναι ένα κοινό δικαίωμα για όλους. Δίχως άλλο η ιατρική έχει προοδεύσει παράλληλο όμως συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν επιδημίες, ότι υπάρχουν έκτακτες περιπτώσεις. Υπάρχει αντίσταση, αντοχή, αντίσταση στα αντιβιωτικά. αλλά και πολλές δυσκολίες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ε, γυναίκε και τα παιδιά που πολλέ φορέ υποσυτίζονται ή ζουν σε κατάσταση ένδυα. Η δική σα μαρτυρία ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, κυρίω όταν μα μιλήσατε για το έργο όλων αυτών που εργάζονται στην ε, ΠΟΗ σε όλο τον κόσμο. Μπράβο σας, άξιοι, άξιοι όλοι σας. Πιστεύω ότι όλοι μας καταλάβαμε πόσο αφοσιωμένοι είναι οι άνθρωποι ε, που δουλεύουν στην οργάνωσή σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συλλογικά είναι οι πρώτοι που δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια στον κόσμο. Αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερη ευθύνη για μας και η εβδομάδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια καλή ευκαιρία για το θυμηθούμε. Μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Η κατάσταση ε, συνεχίζει να ε, παρουσιάζει πολλές ανισότητες, όπως έδειξε η τελευταία έκθεση για την υγεία στην Ευρώπη, και ε, ε, υπάρχει η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά υπάρχει και άνεση πρόσβαση. Το δικαίωμα στην υγεία απειλείται ακόμα και σε αυτή την Ήπειρο από ανισότητες ε, διαρθρωτικές κοινωνικού χαρακτήρα. Μπορούμε να αναφερθούμε στην εξάρτηση από το τσιγάρο, από το αλκοόλ και σε θέματα που αφορούν το ε, περιβάλλον. Θίξατε συγκεκριμένα θέματα. Φέρετε ότι η έκταση για την υγεία στην Ευρώπη δεν δίνει όλη τη διάσταση που θα επιθυμούσε να δώσει στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, σκέφτομαι την ατμοσφαιρική ρήπανση που είναι πραγματικό πρόβλημα δημόσιας υγείας είδα ότι μία Γαλλίδα ερευνήτρια βρήκε μία τεχνική που επιτρέπει να εντοπίσει κανείς σωματίδια στο αίμα και στα ούρα, έκανε μελέτες στα παιδιά που ζουν κοντά σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους και διαπιστώνουμε ότι η παρουσία αυτών των σωματιδίων στα ούρα των παιδιών είναι πολύ πιο υψηλή αν τη συγκρίνουμε με παιδιά που ζουν μακριά από έναν οδικό άξονα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όπω τα άλλα. Δεν υπάρχει μόνο η ατμοσφαιρική ρήπανση, υπάρχει η ρήπανση των υδάτων, των εδαφών. Όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα δημόσια υγεία. Η ΠΟΗ λαμβάνει υπόψη τη αυτά τα θέματα, έχει συγκεκριμένου δείκτε προκειμένου να εξετάσει την επίπτωση που έχουν όλα αυτά στην υγεία. Από την άλλη, η παχυσαρκία σαφώς, σαφώς θεωρείται ως μία καλπάζουσα απειλή σε ό,τι φορά το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων. Το ΠΟΗ θεωρεί την παχυσαρπία χρόνια ε, ασθένεια. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να θεωρηθεί χρόνια ασθένεια. Στην περίπτωση αυτή, ποιε είναι οι συστάσεις για την καταπολέμηση αυτής της επιδημίας παχυσαρκία. Τρίτο σημείο, μας μιλήσατε για τα εμβόλια. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάλυψη, αλλά και εκεί υπάρχουν ανισότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα βρέφη. Και αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα επιθυμούσα να γνωρίζω τι κάνει η οργάνωσή σας για να καταπολεμήσει την ε, καχυποψία που υπάρχει για τα εμβόλια και η καχυποψία αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι κάνει λοιπόν ε, η ΠΟΗ για να διευκολύνει την πρόσβαση στα εμβόλια σε χώρες που αυτό δεν θεωρείται δεδομένο. Σας ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρόστετ. Να ακούσουμε μερικές ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Όπως θέλετε, εσείς το, το αφεντικό. Παρακαλώ, παρακαλώ, να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή της ΠΟΗ ε, και να σας πω ότι μας ενέπνευσε πολύ η ομιλία σας. Δυστυχώς κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την επέτειο ε, της επίθεση στο Βούκοβαρ ε, στα πλαίσια του πολέμου που έγινε στην πρώην Ιουκοσλαβία πριν από 27 χρόνια. Γι' αυτό δυστυχώς δεν θα παραμείνω για να ακούσω τι ε, απαντήσεις Θα με ενημερώσει όμως ε, η βοηθός μου. Η ψηλή τιμή των φαρμάκων είναι μεγάλο πρόβλημα σε πολλές χώρες ε, και είναι γενικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας από τους παράγοντες που ε, απειλεί την βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας η ψηλή τιμή των φαρμάκων. Πολύ συχνά συζητήσαμε για το θέμα αυτό στο παγκόσμιο προσκήνιο, σαν είναι πρόβλημα μόνο των τρίτο ήταν μία ενεπτυγμένων πρόβλημα, είτε των μη ανεπτυγμένων χωρών. Κι όμως, εγώ προέρχομαι από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υψηλές τιμές φαρμάκων. Και αν λάβουμε υπόψη την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ε, τις ώρες αποκατάστασης και την απώλεια ωρών εργασίας, το κόστος είναι τεράστιο. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τις αρμοδιότητες θα πρέπει να προωθήσει κάποια βήματα και κάποιες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται διαφάνεια σε πολλούς τομείς, κυρίως για τις δράσεις της φαρμακοβιομηχανίας και των εθνικών συστημάτων υγείας. Τα τελευταία 20 χρόνια ε, οι τιμές κάποιων φαρμάκων έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που οι πολίτες πια δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακα, κάτι που επίσης ε, απειλεί τη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων υγείας μας. Και σίγουρα με τη γύρεση του πληθυσμού το πρόβλημα θα επιδεινωθεί και με την επέλαση των καρκίνων στο μέλλον θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προωθήσουμε τα καινοτόμα φάρμακα και να μην αποθαρρύνουμε τους φαρμακοβιομήχανους να επενδύσουν στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ευχαριστώ. Thank you Ωραία. Θέλετε να απαντήσετε στι δύο αυτές παρεμβάσει. και μετά θα συνεχίσουμε το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Καταρχά, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, οι θέσει μας με το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου ταυτίζονται. Το θέμα της υγείας είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτοσκοπός και γι' αυτό το λόγο υπάρχει στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από 70 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν το εφαρμόζουμε αυτό με πολιτική δέσμευση. Όπως πολύ σωστά είπατε, μία από τις προκλήσεις στην Ευρώπη Βεβαίω, η Ευρώπη είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. Ε, το θέμα της ισότητας συνεχίζει να είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα και το τόνισα και στην ομιλία μου και αυτό ήταν ε, εξάλλου ένα από τα ευρήματα που ήδη συζητήσαμε. Στην ουσία λέμε το ίδιο πράγμα. Σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένου τομεί που αναφέρατε, η ρήπανση του αέρα για παράδειγμα, η ΠΟΗ οργάνωσε την πρώτη διάσκεψη για τη ρήπανση του αέρα. Η ρήπανση του αέρα τίθεται ως θέμα που έχει σχέση με το περιβάλλον, όχι με την επίπτωση που έχει στη υγεία των παιδιών και των ελληνικών. Όπως γνωρίζετε, επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά. Πολλά παιδιά παρουσιάζουν άσθμα και όταν εκτεθούν σε πολύ μεγάλη ε, ρήπανση του αέρα, ενδεχομένως θα προκύψουν επιπτώσεις για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού. Όλα αυτά βεβαίως είναι τεκμηριωμένα που σας λέω. Όχι μόνο αυτό. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο και καρδιαγκιακά νοσήματα. Αυτό είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ότι η ρήπανση του αέρα είναι κακή για την ανθρώπινη υγεία. Σε πολλές χώρες πετάμε ό,τι βρώμικο στον αέρα. Είναι σαν να τα πετάμε στο νερό που αρχίζει να έχει μία αποφορά και να ε, μολύνεται. Δεν το βλέπουμε, αλλά όπως είπατε και εσείς, έχουμε ε, προσωμιωτές που δείχνουν το επίπεδο ρήπανση σε πολλές πόλεις και το επίπεδο ρήπανση είναι πραγματικά επικίνδυνο σε πολλές πόλεις. Και έχουμε τα πρότυπα ποιότητα του αέρα της ε, ΠΟΗ που ε, δεν έχουν καμία σχέση με τα πρότυπα της ποιότητας του αέρα. Πραγματικά θα ήθελα να τονίσω αυτό το θεματολόγιο και θα ήθελα να τύχουν αυτά τα θέματα της απαιτούμενης προσοχής ε, στις συζητήσεις με τα μέλη της Επιτροπής ε, σήμερα. Αναφερθήκαμε στο θέμα των συμβάσεων για την ποιότητα του αέρα ε, όπως για παράδειγμα η σύμβαση FCTC για τον ε, ε, καπνό. Όσο ανεχόμαστε αυτό το επίπεδο καταστροφής για την ανθρώπινη υγεία, τόσο τα πράγματα παραμένουν έτσι. Υπάρχουν συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και τις συζητήσαμε και με τα μέλη της Επιτροπής. Θα θέλαμε εσείς να γίνετε η δική μας φωνή. Γιατί η φωνή αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε δεσμευτικές συμβάσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπνέουν καθαρότερο αέρα. Η ποιότητα του αέρα, ο καθαρός αέρας είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο αέρας που αναπνέουμε δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνος. Ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή μας. Και βεβαίως αυτό έχει σχέση και με την ρήπανση των υδάτων λοιπά. Μιλάμε εδώ για ένα καθαρό περιβάλλον από όλε τι απόψει. Μιλάμε και για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τα χημικά προϊόντα. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό και βέβαια η ρήπανση του αέρα είναι θέμα σημαντικό. Η παχυσαρκία δεν θεωρείται χρόνιο νόσημα, αλλά ως, επικίνδυ, ως επιβαρυντικός παράγοντας και θα πρέπει να θεωρηθεί ως τέτοιος. Σε ορισμένες χώρες είδα έναν επικίνδυνο συνδυασμό. Ο αριθμός των καπνιστών είναι πάρα πολύ ψηλό, 40%. Ας πούμε οι ε, ε, άνδρες ενήλικες. Επίσης ψηλό ποσοστό παρουσιάζει παχυσαρκία. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που οδηγεί σε πρόωρο θάνατο. Και όλα αυτά, σε όλα αυτά προστίθεται και η κατάχρηση του ινοπνεύματος. Έλλειψη φυσικής γυμναστικής, υνοπνεύμα, ε, κάπνισμα και Τέλος, ακατάλληλη διατροφή θα μπορούσε να είναι οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν ε, την, τον επιπολασμό των το μη ε, λιμωδών νόσων. Ο, οι επιβαρυντικοί παράγοντες πίσω από αυτές τις μη λιμώδεις νόσους είναι αυτοί αυτή που ανέφερα πέρα από άλλους που είναι η ρήπανση του αέρα. Η ρήπανση του αέρα σκοτώνει 7 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο. Είναι μία από τις βασικές αιτίε πρόωρου θανάτου. Η υπαχυσαρχή αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντο και θα πρέπει να αντιμεστώ ε, αντιμετωπιστεί. Στην ΠΟΕ έχουμε μία επιτροπή, ειδική επιτροπή και ο αγώνας μας έχει μετατεθεί ε, σε ένα άλλο επίπεδο. Γιατί πραγματικά πρόκειται για έναν κίνδυνο, για μια πρόκληση για όλο τον ε, κόσμο. Γιατί πλήττει όλες τις χώρες, τις χώρες ε, τις πλούσιες και τις στοχεύει τον ίδιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη εμβολιασμού αφορούν και την Ευρώπη από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018. Το ξέρετε ότι υπήρξαν πάνω από 60.000 περιπτώσεις οτίτιδας στην ε, ε, Ευρώπη. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Πώς είναι δυνατόν για την Ευρώπη να χάνονται παιδιά από μια τέτοια νόσο. Εδώ μιλάμε για χώρες μέλη της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη βοήθεια των εμβολίων με την ευλογιά. Είμαστε στα πρόθυρα του να εκριζώσουμε την πολιομιελίτιδα. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σημαντικά λόγω των εμβολίων. Τα παιδιά αναπτύσσονται και φτάνουν στην ενήλικο ζωή λόγω των εμβολίων. Καρπορεμάμε στο Κονγκό την, τον έμπολα καλύτερα λόγω των εμβολίων. Πάνω από 32.000 άνθρωποι εμβολιάστηκαν. Ε, αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια, από τους 32.000 που εμβολιάστηκαν, το ένα τρίτο από αυτούς θα είχαν παρουσιάσει την ε, ε, νόσο έμπολα. Τα, ε, οι περιπτώσεις θα είχαν φτάσει 10.000 και παραπάνω. Η, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα εμβό, τον εμβολιασμό, την αξία του εμβολιασμού. Κάποιος σε κάποιο μέρος του κόσμου μεταδίδει μια ψευδή είδηση και αυτό αμφισβητεί τα ωφέλη τον ε, του εμβολιασμού. Στα χέρια σας είναι να πείτε φτάνει ως εδώ. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά. Ο εμβολιασμός βοήθησε και μας και τα παιδιά μας για πολλά χρόνια. Και συνεχίζουν να βοηθάνε και θα το κάνουν στο Δινεκές. Είναι επικίνδυνο να αμφισβητούνται τα, ε, να αμφισβητεί το εμβολιασμό. Ε, αυτή η αμφισβήτηση μας ε, επαναφέρει στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Είναι επικίνδυνο. Ε, έθεσε ένα θέμα ο συνάδελφος ε, για την αντιμικροβιακή αντοχή. Αν μπορεί να προλάβει κανείς μία νόσο, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί αντιβιωτικά ή φάρμακα, είστε στη διαδικασία πρόληψης. Δεν, ε, ε, δεν εμφανίζεται η νόσος. Συνεπώς, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος, χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη. Υπάρχουν πάρα πολλές λανθασμένες ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά γίνονται αποδεκτά από μεμονωμένα άτομα και από οικογένειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των φαρμάκων, σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, διότι δεν γίνεται να υπάρξει καθολική κάλυψη υγείας χωρίς πρόσβαση σε προσιτά ποιοτικά φάρμακα. Αυτό έχει προτείνει και το πάνελ και ο Γενικός ε, Γραμματέας. Αυτό που μένει είναι να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις. Και φυσικά να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και να μην παραμερίζεται ε, το θέμα της καινοτομία. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω πως μπορεί να επιτευχθεί μια ισορροπία, όμως χρειάζεται να καθοριστεί από την αρχή, να επαναπροσδιοριστεί και να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της πρόσβασης στα φάρμακα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε καθολική πρόσβαση ε, στα φάρμακα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Κέκα. Ο κύριος Πιέχα. Θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας που έχει την καλοσύνη να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναμφίβολα, η 70η επέτειος από την ίδρυση της ΠΟΗ είναι εξαιρετική ευκαιρία για να ε, συγχαρούμε αλλά και να ευχαριστήσουμε την ΠΟΕ γιατί είναι σημαντικό στοιχείο για την παγκόσμια υγεία. και φυσικά θέλουμε ισότιμη πρόσβαση σε προσιτής υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πολύ σημαντική επίση είναι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο είδωρο και σε καλέ, καλές υγειονομικές συνθήκες, σε υγιείς συνθήκες απασχόλησης. το δικαίωμα στο καλό και υγιές περιβάλλον. Και πολύ σημαντική είναι η πρόσβαση του κόσμου στην πληροφόρηση και στην διαπαιδαγώγηση για την υγεία. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Και σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι η βάση της δημόσιας υγείας. Και η υγειονομική περιθαλψή είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα, αλλά όχι το μοναδικό ε, το παραδικό σκέλος υγείας και σίγουρα είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε την υγεία ως δικαίωμα και μάλιστα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, το δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώνεται στον καταστατικό χάρτη, στο σύνταγμα της χώρας. Γι' αυτό το κράτος, ο κρατικός μηχανισμός οφείλει και εξαναγκάζεται λόγω της κατοχήρησης του συντάγματος να εξασφαλίσει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στα συναφή δικαιώματα που σχετίζονται με την πρόθεση της υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, ασχολείται με αυτά τα θέματα και έχει εκδώσει πολλές συστάσεις και έγγραφα που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται παρόλο που αποτελεί υποχρέωση των κυβερνώντων και πραγματικά είναι θεμελιώδες δικαίωμα για την ε, διαμόρφωση μιας ευημερία και ε, θετικών ε, βιωτικών συνθήκων. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους πρώτους δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας και έχει τεράστιο δυναμικό και μάλιστα το δυναμικό της βρίσκεται σε διάφορους οργανισμούς, τον Οργανισμό Φαρμάκων, του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, Ελέγχου των Επιδημιών. Και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας καλό θα ήταν να έχει πολύ στενό και τακτικό διάλογο με όλους αυτούς τους οργανισμούς και φυσικά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρόλαβα να διαβάσω ακόμη ε, διεξοδικά αυτό το παγκόσμιο σχέδιο δράσης ε, για την ε, υγεία για όλους, αλλά θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο, ανεκτήμητο θα έλεγα έγγραφο και ε, σας διαβεβαιώ ότι και η πολιτική ομάδα αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσσωμα θα στηρίξει την πρωτοβουλία του ΠΟΗ. Και μια πιο δύσκολη ερώτηση που ίσως δεν πληρεί αυτόν τον ερωταστικό χαρακτήρα της 70ης επαιτίου. Θα ήθελα να ενημερωθώ για κάποια θέματα που κατά τη γνώμη είναι σημαντικά. Η ΠΟΗ έχει κάποιο γενικό σχέδιο για την κατάλληλη προετοιμασία και πρόσβαση ε, στα, στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, γιατί υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όχι μόνο στις χώρες Αφρικής, αλλά ακόμη και στην Ευρώπη. Ε, χωρίς όμως ε, ιατρικά στελέχη, πώς να μιλήσουμε για διαπαιδαγώγη σωστή και για να μιλήσω για περίθαλψη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε μια κατάρτιση σε στελέχη στον ιατρικό κλάδο παγκοσμίω, γιατί υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Και ένα άλλο θέμα, πολύ λεπτό, αφορά την παρηγορητική αγωγή. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και μερικές φορές δημιουργεί κάποια εδώ. Κι όμως ο θάνατο είναι κάτι το σίγουρο, το βέβαιο. Ο αξιοπρεπή θάνατο όμω δεν είναι τόσο σίγουρο και βέβαιο. Και το θέμα τη παρηγορητικής αγωγή είναι πολύ ευαίσθητο και δύσκολο. Ασχολείστε με το θέμα αυτό, θα προτείνετε κάποιε διαδικασίε, κάποιε μεθόδου, ώστε να εξασφαλίσουμε χάρη στην παρηγορητική αγωγή έναν αξιοπρεπή θάνατο που δεν είναι, πια, που δεν είναι δυστυχώς κάτι δεδομένο. Επίσης, κατά την μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ένα από τα καινούργια στοιχεία θα πρέπει να είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι ένα σύνθημα, μια εποδός που επανέρχεται πολύ συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε συζήτηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο προπολογισμό τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Από ό,τι ξέρω είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια ο προπολογισμό ε, τη Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγεία. Και η κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού δεν γίνεται κατά ανάγκη με μεγάλη διαφάνεια. Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν την κατανομή του προϋπολογισμού ε, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση των ε, ε, υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο στις χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη. Και το λέω αυτό για το Μεξικό, που εκεί αναφυσβήτητα κάποια θέματα σε ό,τι αφορά το ύψος των κονδυλίων. Και εκεί δυστυχώς δεν ε, πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις της διαφάνειας. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ θερμά για την ομιλία σας και σας διαβεβαιώ ότι ε, θα στηρίξω πλήρως το παγκόσμιο σχέδιο δράσης, ώστε η ζωή των κατοίκων αυτού του πλανήτη να είναι αξιοπρεπής και καλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιέχα. Κυρία Μάισνερ, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Γενική Διευθυντή, βρίσκεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα και εγώ να χρησιμοποιήσω τη δική μου γλώσσα, τα γερμανικά, για να σα ευχαριστήσω εξ ονόματο των φιλελευθέρων ε, που ήρθατε. Κρίμα που δεν είναι ακόμα περισσότεροι ευρωβουλευτέ εδώ, διότι θα θέλαμε πραγματικά να ε, σας ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον ε, Λίσαντα. Θεωρώ πω το παγκόσμιο σχέδιο δράση είναι πολύ καλό. Χαίρομαι πολύ που έχουμε και το βιβλιαράκι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Ε, να είστε σίγουρος πως θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για καλή συνεργασία. Κάποιες ερωτήσεις, ε, γιατί ακούστηκαν ήδη πολλέ, Καταρχάς, ε, για την πλατφόρμα Right to Health, δικαίωμα στην υγεία. Υπάρχει κάποια οικονομική στήριξη, κάποιοι χορηγοί ε, ποιος είναι ο προϋπολογισμός της πλατφόρμας και πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια. Μετά, Αναφερθήκατε σε ορισμένες ασθένειες τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα. Υπάρχουν όμως και άλλες. Υπάρχουν πνευματι... Υπάρχει το θέμα της πνευματικής ε, υγείας. Έχετε ε, αυτές ε, τις ασθένειες κατά νου. Υπάρχουν και άλλες. Μετά, τι γίνεται με το HIV είναι μία νόσος ε, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ε, ικανοποιητικά. Υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση στην έρευνα. Εσείς ε, τι κάνετε για να καταπολεμήσετε την εξάπλωση του UHIV στην Αφρική. Και τελευταία ερώτηση που αφορά κυρίως την Αφρικανική Ήπειρο. Ο τι κάνει για να καταπολεμήσει και να εξαλείψει τον ακροτηριασμό των ε, γεννητικών οργάνων. Είναι μία μάστιγα πραγματικά και σίγουρα το δικαίωμα στην υγεία αφορά και αυτό. Αυτά ήταν οι ερωτήσεις από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Πέτερλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια και για την παρουσίαση του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης. Μιλώ και εξ ονόματος ε, όσων είναι ταγμένοι στη μάχη κατά του καρκίνου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις τελευταίες δεκαετίες παρά την πρόοδο της ιατρικής ε, ο καρκίνος παραμένει τεράστια πρόκληση όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα. Αναφέρατε κάποιους δείκτες σχετικά με αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία διαγράφονται οι αρχές ε, για όλες τις πολιτικές. Και αναφερθήκατε επίσης στις ανισότητες ή μάλλον τις διαφορές που υπάρχουν εδώ. Το κόστος των φαρμάκων και της ε, θεραπείας αυξάνεται επικίνδυνα και αυτό θα καταστήσει δύσκολη την εφαρμογή της αρχής αυτής ε, της καθολικής ε, κάλυψης για όλους τους ασθενείς. Προσωπικά καλωσορίζω το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Υγεία και για μένα λέξη κλειδί είναι η επιτάχυνση. Νομίζω πως ε, δεν υπάρχει ανάγκη να καινοτομήσουμε σε πολλούς τομείς, ε, διότι έχουμε γνώση και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε αρκετέ γνώσεις έτσι ώστε να γίνουμε ταχύτεροι στην αντιμετώπιση ασθενειών. Και ε, να σας αναφέρω ότι έγινε χθε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ήταν εκεί ο David Beasley, εκτελεστικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος και αναφέρθηκε στη ζώνη του Σαχέλ, όπου χρησιμοποιείται ένα επιστημιστικό πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους πάρα πολύ παλιές, πάνω από εκατοντάδων ετών. Φυτεύουν δέντρα στη ζώνη του Σαχέλ, προσπαθούν να σταματήσουν την ε, εξάπλωση της ερήμου Φαντάζομαι γνωρίζετε γι' αυτό. Και η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως ημισέλληνος. Ίσως τη γνωρίζετε μια και είστε από την Αιθιοπία. Είναι μια πάρα πολύ απλή μέθοδος, η οποία όμως είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και νομίζω πως και σε άλλους τομείς μπορούμε να δράσουμε με τρόπο πιο συνεκτικό και ολοκληρωμένο. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Λοιπόν, και θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την στρατηγική για ε, την παραδοσιακή ιατρική του ΠΟΗ. Οι ασθενείς δέχονται μόνο ένα φάρμακο και αυτό είναι το φάρμακο που τους γιατρεύει. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα καλύτερα από την παραδοσιακή ιατρική και τη σύγχρονη ιατρική και ας αφήσουμε κατά μέρος τις ιδεολογικές διαμάχες για το ποιο φάρμακο είναι καλύτερο. Πιστεύω πως ε, αυτό θα χαροποιήσει όλους τους ασθενείς, όταν δηλαδή ξεφορτωθούμε αυτές τις ε, ιδεολογικές προσεγγίσεις και υιοθετήσουμε την αρχή της αποτελεσματικότητας, διότι αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος πάλι σε εσά, δόκτωρα Τέντρος. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα που επισημάνατε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πιέχα ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις αιτίε του προβλήματος ό,τι αφορά αυτό το δικαίωμα στην υγεία. Και αν φροντίσουμε τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε και το περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε, θα λύσουμε το πρόβλημα της υγείας. Γιατί ε, τα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από τους παράγοντες κινδύνου που βλέπουμε σε αυτούς τους τομείς. Οπότε θα πρέπει να δούμε τα αίτια ε, που υποσκάπτουν την υγεία. Και σίγουρα ε, το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης περιέχει ε, τρεις ε, προτεραιότητες στρατηγικές. Καταρχήν, καθολική κάλυψη υγείας. Δεύτερον, ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τα έκτακτα περιστατικά, δηλαδή ασφάλεια. Και το τρίτο είναι υγιής πληθυσμοί, δηλαδή ποιοι είναι οι παράγοντες που πειράζουν την υγεία. Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένας από αυτούς, όλα αυτά που μας είπατε. Και το να κρατήσουμε τον κόσμο υγιή, να προλάβουμε την αρρώστια. Γιατί να παραπέμπουμε κάποιους στα νοσοκομεία ή στην υγειονομική περίθαλψη, αυτό είναι ένδειξη ήτας, γιατί το κακό έχει γίνει. Να προλάβουμε είναι το θέμα, να προλάβουμε την ε, εμφάνιση της, της νόσου, της ασθένειας, αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες που επιδεινώνουν την υγεία και αποτρέποντας την εμφάνιση των νόσων. Και αυτό οργανώνομαστε και ε, από τους πυλώνες που έχουμε στις στρατηγικές μας, ε, ένας βασικός παράγοντας στρατηγικής είναι ο υγιής πληθυσμός. Να κρατήσουμε τον κόσμο υγιή, γερό, να μην φτάσουμε στην αρρώστια. Γι' αυτό το λέει το έγγραφο. Και δεν θα πρέπει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να είναι ε, η οργάνωση που θεραπεύει αρρώστους. Δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός. Ο προσανατολισμός μας είναι να κρατήσει υγιείς τους ανθρώπους σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρου του παγκόσμιου σχεδίου. Όντως, ε, υπάρχει έλλειμμα στο εργατικό δυναμικό του κλάδου υγείας. Έχουμε ένα έλλειμμα 18 εκατομμυρίων ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τεράστιος αριθμός. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό με καινοτόμου τρόπου και καινοτόμε ιδέε. Και αυτό θα είναι ένα τμήμα τη Παγκόσμια Στρατηγική που θα ε, σχεδιάσουμε και θα αντιμετωπίσουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη ε, το κενό αυτό, το έλλειμμα των 18 εκατομμυρίων ε, εργαζομένων στον κλάδο της υγείας. Πάντως, έχουμε ήδη κινητοποιηθεί για να καλύψουμε αυτό το κενό. Σε ό,τι αφορά την παρηγορητική, ανακουφιστική αγωγή, υιοθετούμε την προσέγγιση της υγείας από τη μήτρα στον τάφο, όλη τη διάρκεια της υγείας. Δηλαδή, προωθούμε την υγεία, αποτρέπουμε τις ασθένειες, προλαμβάνουμε, ε, θεραπεύουμε, ε, θεραπεύουμε κάποιον, προσφέρουμε θεραπευτική αγωγή, αποκατάσταση αν χρειάζεται και μετά παρηγορητική αγωγή. Θα πρέπει να καλύπτουμε όλο το φάσμα όταν μιλούμε για τις υπηρεσίες υγείας. Όλη τη διάρκεια ζωής, όλα τα βήματα και γι' αυτό υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση της πορείας της ζωής από τη μήτρα στον τάφο. Και ευθυγραμμίζομαι πλήρως με αυτά που μας είπατε για τους πόρους. Ο προϋπολογισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι 2,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. 4,5 δισεκατομμύρια διετία. 2,4 το έτος δισεκατομμύρια. Είναι μικρός ο προϋπολογισμός. 2,5 εκατομμύρια σε μερικές χώρες υψηλού εισοδήματος είναι προϋπολογισμός ενός νοσοκομείου. Και σίγουρα δεν είναι μεγάλος ο προϋπολογισμός της ΠΟΗ και ευχαριστούμε βέβαια τους δωρητές μας, ε, τους εταίρους μας για τη γενοδορία τους. Πάντως όποιος και είναι ο προπολογισμό της ΠΟΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά, συνετά, αποτελεσματικά, να πιάνει τόπο. Και ε, χρησιμοποιούμε τους πόρους μας, τα κονδύλια μας, σε βάση των προτεραιοτήτων μας. Αυτό κάνουμε. Και όταν ε, λέω βάση των προτεραιοτήτων εννοώ ε, βλέπουμε ποιες προτεραιότητες θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, τις περισσότερες συνέπειες ε, για τον κόσμο. Και έτσι κινούμαστε. Επίσης έχουμε συστήματα εσωτερικής αξιολόγησης. Τώρα θα περάσουμε και στην εξωτερική αξιολόγηση και ένα συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Έτσι θα δούμε πώς υλοποιούμε τους στόχους μας και πώς χρησιμοποιούμε και τους πόρους μας. Και γι' αυτό είναι σημαντική και η εξωτερική αξιολόγηση για να μας βοηθήσει να δούμε κάτι που ίσως χάνουμε όταν τα βλέπουμε εκ των έσω. Όταν είναι κανείς πολύ κοντά δεν βλέπει καλά την κατάσταση και κάποιος που βλέπει από απόσταση τον βοηθάει να δει καλύτερα τα πράγματα. Οπότε ό,τι αδυναμίες και αν αντοπίσουμε, είμαστε ανοιχτοί και θα τις αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία, καλύπτει και την άνοια αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας. και έχουμε προτεραιότητα το καρκίνο, το διαβήτη, ε, χρόνιες πνευμονοπάθειες. Αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότητες. Αλλά τώρα προσθέτουμε και την ψυχική υγεία στις προτεραιότητές μας. Οπότε έχουμε καρδιακά νοσήματα, καρκίνο, πνευμονοπάθειες και το διαβήτη και μετά έχουμε την ψυχική υγεία ως βασική προτεραιότητα. Η ψυχική υγεία και ένα από τα προβλήματα σε πολλές χώρες είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες ή δεν υπάρχουν παντού. Μόνο σε ειδικευμένα ιδρύματα παρέχονται ή σε νοσοκομεία. Και μερικέ φορέ αντιμετωπίζουμε του ψυχικά νοσούντε ω εγκληματίε, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Η ψυχική υγεία και τα προβλήματα τη ψυχική υγεία είναι ε, σαν οποιαδήποτε άλλη αρρώστια. Κάποιο μπορεί να έχει στομαχόπονο, άλλο μπορεί να έχει μια ψυχική νόσο. Είναι μια κανονική ασθένεια και η ψυχική νόσος και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Κάποιες όμως οικογένειες αντιμετωπίζουν ακόμα και τα παιδιά τους ως εγκληματίες και υπάρχει το στίγμα της ψυχικής νόσου που ξεκινάει στην οικογένεια. Το πρόβλημα με την ψυχική υγεία είναι το στίγμα στον τομέα της υγείας, στα ιδρύματα, αλλά και το στίγμα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θέλουμε να αυξήσουμε την επαγρύπνηση της κοινωνίας και να αντιμετωπίσει την ψυχική υγεία ως ένα κοινό πρόβλημα υγείας και να το συνεκτιμήσουμε στο σύστημα υγείας, ακόμη και στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ώστε να μην αντιμετωπίζεται η ψυχική υγεία ως ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά ενό κοινό πρόβλημα υγείας που θα περιλαμβάνεται σε όλο το σύστημα και στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Και κανένα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγκληματία όταν νοσεί ψυχικά. Αυτός αυτή είναι η προώθηση λοιπόν του θέματος. Επίσης, ε, η Άννη είναι τμήμα της ψυχικής υγείας οι διαστάσεις είναι τεράστιες εδώ. Και όσοι νοσούν από άνοια στιγματίζονται και από τις ίδιες οικογένειές τους μερικές φορές. Και πραγματικά οι διαστάσει του προβλήματο είναι μεγάλες. Και όταν λέω ψυχική υγεία περιλαμβάνω και την άνοια. Είναι σφαιρική η προσέγγιση. Και υπάρχει δέσμευση και μάλιστα πολλές χώρες πρωτοστατούν στα θέματα αυτά, μερικές και ευρωπαϊκές και ο Γενικός Γραμματέας είναι ιδιαίτερα προσιλωμένος στο ζήτημα της ψυχικής υγείας και πραγματικά και εμείς στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα προωθήσουμε αυτά τα θέματα και χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια ώστε να δημιουργήσουμε μια όθηση και πρόσφαρες προϋποθέσεις για να αυξήσουμε την επαγρύπνηση, γιατί η ψυχική υγεία είναι ένας ύπουλος και σιωπηλός δολοφόνος που μερικές φορές ε, τον παραμελούμε και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ό,τι αφορά το AIDS, η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του ιού του AIDS ε, ε, έχει αρχίσει να μειώνεται. Γενικώ ό,τι αφορά τον ιό HIV έχουμε αρκετή επιτυχία. Μειώνεται η, η επιδημία του AIDS σημαντικό επίτευγμα και η θνησιμότητα ε, του AIDS στο παρελθόν ήταν πολύ υψηλή. Και ιδιαίτερα σε μερικές μικρές ε, πόλεις που όλοι γνωρίζουν τους πάντες, βλέπουμε ποιο είναι το εύρος ε, των κρουσμάτων και των θανάτων λόγω AIDS. Και πολλές οικογένειες αποδεκατίστηκαν και απελπίστηκαν. Και όταν μια οικογένεια απελπίζεται, το έθνος κλονίζεται, γιατί η οικογένεια είναι ο πυλώνας της ελπίδας ενός έθνους. Έτσι ε, ξεκινήσαμε μία αναβάθμιση της πρόληψης αλλά και της, περιθα... και της περιθαλψής 21 εκατομμύρια ε, ε, υπόκειται σε θεραπεία και έχει μειωθεί κατακόρυφα η θνησιμότητα λόγω AIDS και αυτό δίνει και πάλι ελπίδα στις οικογένειες οπότε η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά για το AIDS και αυτό είναι ένα από τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την παγκόσμια αλληλεγγύη ε, για να καταπολεμήσουμε μια σημαντική νόσο που επηρεάζει πολλές χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να χάσει το χαρακτηρισμό της επιδημίας του AIDS και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη. Και παρόλο που γενικώ υπάρχει μείωση του AIDS, σε μερικές χώρες υπάρχει αύξηση. Θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε τις δράσεις μας και να αντιμετωπίσουμε μια για πάντα το θέμα. Σε ό,τι αφορά τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, είναι ένα πρόβλημα υγείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και θέμα δικαιωμάτων, όπως είπατε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί οι λοιμώξεις μεταδίδονται λόγω αυτής της κακής πρακτικής, όχι μόνο του ακροτηριασμού γεννητικών οργάνων που ε, επηρεάζει τη ζωή, ολόκληρη τη ζωή όλων των κορισιών που ε, υπόκειται σε αυτή, αλλά μπορούν λόγω μόλυνση πολλά κορίτσια να χάσουν και τη ζωή τους τη διάρκεια της επέμβαση. Οπότε θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το θέμα, γιατί προκαλεί πρόβλημα όχι μόνο στην υγεία, αλλά και γενικό και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή ιατρική, και για την εμπειρία στο Σαχέλ, την ημισέλινο, είχα προσωπική πείρα και μάλιστα συμμετείχα στη, στην πρωτοβουλία αυτή για να βελτιώσουμε την οικολογική κατάσταση μερικών περιοχών στην Αιθιοπία και το είδα και με τα μάτια μου ε, όταν χρησιμοποίησαμε την ημισέλη, όταν επανήλθε η βλάστηση και πώς βελτιώθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και όταν άρχισε το όλο περιβάλλον να βελτιώνεται και λόγω της βελτίωσης και του, των υπόγειων υδάτων ε, μπορέσαμε να αρδεύσουμε και όλα μερικά χωράφια και με την ε, άρδευση η παραγωγικότητα της γεωργίας βελτιώθηκε, οπότε είχαμε βελτίωση στο περιβάλλον και βελτίωση στο αγροτικό εισόδημα με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και είναι μια τεχνολογία αυτή που είναι γνωστή αιώνε ολόκληρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ακόμη και σήμερα. Τι χρειάζεται? Δεν χρειάζεται καν πολλά χρήματα. Αν πείσουμε τους γεωργούς, ε, είναι δική τους δουλειά. Και μάλιστα είναι δωρεάν ώρες απασχόλησης και αν είναι πρόθυμοι και πιστούν οι γεωργοί να βάλουν το μόχθο τους σε αυτή την προσπάθεια, θα τα καταφέρουμε. Η ιστορία μας έχει διδάξει πολλά θετικά παραδείγματα. Και υπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες, πρακτικές, ιδέες που μπορεί να ξεκίνησαν στο παρελθόν, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα, ακόμη και για τον τομέα υγείας. Και εκτός του ελέγχου των πρακτικών που έχουμε και τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τώρα στον τομέα υγείας, σίγουρα σημαντικές θα είναι και οι επενδύσεις στην ψηφιακή υγεία. Γιατί το μέλλον της υγείας θα επηρεαστεί φυσικά από την ψηφιακή υγεία. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Και εμείς τώρα στην ΠΟΗ θέλουμε να πρωτοστατήσουμε, να είμαστε διορατικοί σε αυτά τα θέματα, να αντιληφθούμε την ψηφιακή, υγεία και τα πλονεκτήματά της και να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος ανθρωπότητας. Η τεχνολογία της ψηφιακής υγείας θα έχει τεράστια επιρροή στην υγεία και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή ιατρική, συμφωνώ και δεν αποκλείεται η παραδοσιακή ιατρική, τη σύγχρονη ιατρική. Μπορούμε να συνδυάσουμε και τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα. Και αυτό κάνουμε στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Δεν αλληλοαποκλείονται οι μέθοδοι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους, όλη τη γνώση, όλες τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στις κοινωνίες μας. Αυτά και σας ευχαριστώ και πάλι. Πολύ χρήσιμες ερωτήσεις, πολύ σημαντικές και βλέπω ε, πόσο ε, προσιλωμένη είστε σε αυτό το θέμα και με χαροποιεί αυτό σας το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε και φίλεν Ντάνκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, Δόκτωρα Τέντρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνήσαμε να υπογράψουμε όλοι μαζί μια κοινή δήλωση η οποία θα εκφράσει την ε, συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού ε, και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αναγνώριση του σημαντικού έργου του ΠΟΗ στην πρόθεση του Παγκοσμίου Σχέδιου Δράσης για την υγεία για όλους. Μπορείτε λοιπόν να την υπογράψετε. Θα μας βοηθήσει και η γραμματεία να έχει την καλοσύνη. Και αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά θα κλείσουμε τη σημερινή συνεδρίαση με ένα ποτήρι σαμπάνιας.